την κυρία Κρούς που θα μας παρουσιάσει ε, τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κλίση e-call. Α, δεν ξέρω για τη μερίσια διάταξη, έχουμε κανένα πρόβλημα, όχι. Θα δώσω μέσα το λόγο στην κυρία Κρούς, η οποία θα μας παρουσιάσει σε 15 λεπτά ε, τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την Ευρωπαϊκή Κλίση e-call. Να δούμε αν έχουν λιανθεί οι τελευταίες δυσκολίες και ξεπεραστεί τα τελευταία εμπόδια και μετά να μιλήσουν οι συντονιστές ένα λεπτό έκαστος έτσι ώστε να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Έχετε το λόγο κυρία Κρούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με επευθύνατε. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερο. Ε, αυτήν την ε, πρόσκλησή σας να παραστώ στην ε, Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσω να μιλήσω όχι μόνο για αυτό το θέμα. Δεν θα εκπλαγείτε φαντάζονται ότι ε, ε οτιδήποτε έχει σχέση με την παλιά μου ζωή παρότι αυτή ήταν τον προηγούμενο αιώνα με ευχαριστεί ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να δούμε πώς ε, τα έξυπνα συστήματα μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν ε, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τους Ευρωπαίους πολίτες. Αναφέρομαι εδώ στο e-call. Γυρνάτε σπίτι σας το βράδυ, το χειμώνα, σαν έναν ευρωπαϊκό δρόμο. Και έχετε ένα πρόβλημα. Και έχετε ένα πρόβλημα και με το αυτοκίνητό σας. Uh, και με το ατύχημα αυτό παγιδεύεστε με κάποιο τρόπο ή λόγω κακών καιρικών συνθήκων ε, και είσαι και ανέστητος. Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι, ε, ε, πόσο σημαντική μάλλον είναι η άμεση ιατρική βοήθεια. Είναι αυτή η golden hour, αυτή η χρυσή ώρα της άμεσης παρέμβασης. Ε, και μπορούν πραγματικά αυτήν την ώρα ε, να σωθούν ζωές και να μην υπάρξουν περαιτέρω και μετέπειτα προβλήματα. Ε, οποτεδήποτε ανιχνευθεί επικίνδυνο ατύχημα τότε οι αισθητήρε αμέσως ειδοποιούν μέσω αυτής της ε, κλίσης και δίνουν πολλά στοιχεία μεταξύ των οποίων και την ακριβή τοποθεσία έτσι ώστε να φτάσουν το δυνατό γρηγορότερο οι βοήθειες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι πλή, είναι, ε, είμαστε πολύ κοντά σε αυτήν την ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το e-call δηλαδή. Και ε, ξέρουμε ότι θα έχουμε και την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Πανευρωπαϊκή Υπηρεσία e-call έχει την δυνατότητα να μειώσει τους θανάτους από ατυχήματα ε, στους δρόμους και να μειώσει κατά τουλάχιστον 6% το κόστος ε, της ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι εάν λειτουργήσει σωστά το e-call θα σώζεται μία ανθρώπινη ζωή κάθε 6 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία έχει ε, ε, εκπονήσει μελέτες έτσι ώστε ε, να υπάρξει καλύτερη δυνατή διευθέτηση και καλύτερη δυνατή εφαρμογή του e-call. Έχουμε σκεφτεί διάφορες περιπτώσεις, ε, αλλά πιστεύουμε ότι η υποχρεωτική εφαρμογή είναι η καλύτερη επιλογή και όσον αφορά την απόδοση κόστους ωφέλους. Γίνεται λοιπόν σύσταση από πλευράς ε, των κρατών, των, της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας να μεταδίδεται το σήμα του e-call η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βεβαίως ε, είναι στρατευμένη στην μείωση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τις χώρες ε, μέλη να βεβαιωθούν και να διασφαλίσουν ότι το e-call σαν υπηρεσία θα μπορέσει να εφαρμοστεί όσο γίνεται γρηγορότερα και σε συνεργασία και σε συνέργεια με το 112 την κλίση αυτόν τον αριθμό θα πρέπει οπωσδήποτε ε, οι ε, ε, operators και οι διάφοροι φορείς των δικτύων να συνεργαστούν πλήρως έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται τα σήματα των e-call μαζί με τα σήματα των επιγουσών κλήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα στείλουμε και ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε όλους τους εμπλεκόμενους ε, ότι μας ενδιαφέρει αυτή η υπηρεσία ε, να αφορά κάθε είδους όχημα και έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είτε είναι αυτοκινητοβιομηχανία είτε είναι κινητά δίκτυα τηλεφωνίας κτλ να δουλέψουν γι' αυτό. Ε, και όσον αφορά το e-call θα κάνουμε μία πρόταση κανονισμού ε, υπό το ευρύτερο, τον ευρύτερο κανονισμό ε, που διέπει τα οχήματα και πάντα μέσα στα πλαίσια της οδηγίας ITS και όπου θα αποσαφηνίζονται τα απαραίτητα στοιχεία του εξοπλισμού που θα πρέπει να έχουν τα οχήματα. Ε, και όσον αφορά τα μη υποχρεωτικά μέρη, βεβαίως ε, ε, συνεργάζονται οι υπηρεσίες μας με τον Αντώνιο Γκατζάνη και με τους άλλους ε, συγγνώμη, με, τους, με τις υπηρεσίες των άλλων δύο συναδέλφων μου επιτρόπων, Ταγιάννη και Ντάλλας και Κάλλας. Και βεβαίως ε, θα συνεχίσουμε την ε, ε, προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει ισομερής εκπροσώπηση όλων των εμπλεκομένων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω των εκπροσώπων τους και των οργανώσεών τους να συνεχίσουμε την εργασία. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει, στηρίζει την ε, ε, ε, τις εκστρατείες ε, ευαισθητοποίησης έτσι ώστε και η κοινή γνώμη ε, να είναι γνώστη των πραγμάτων και επίσης έρχεται σε επαφή με την αντίστοιχη βιομηχανία έτσι ώστε να υπάρχει καλή διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ταυτοχρόνως από τους πολίτες. Το e-call μπορεί να παίξει κατά κάποιο τρόπο και τον ρόλο καταλήτη για άλλες υπηρεσίες όπως είναι ας πούμε τα συστήματα πλοήγησης, ε, η οδική βοήθεια κτλ. Έχουμε δουλέψει για το θέμα αυτό του e-call εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θυμάστε ότι ε, υπήρξε και ένα κονδύλι το οποίο είχε ενταχθεί στην έρευνα για το θέμα αυτό. Ε, εγώ πιστεύω ότι ε, η έρευνα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει να εξευρεθούν λύσεις για προκλήσεις που αφορούν την κοινωνία και που θα βοηθήσουν όλους τους, όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Πολλά έτη εργάζονται οι υπηρεσίες μας έτσι ώστε να καταφέρουν καταφέρουν να συγκεντρωθούν γύρω από ένα τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, έτσι ώστε να βρεθούν συστήματα τα οποία θα είναι απλά, θα μπορούν να λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, να είναι πανευρωπαϊκά ε, ε, συστήματα και τα οποία βεβαίως θα έχουν την δυνατότητα να προσαρμοστούν στην υποδομή των κρατών μελών και βεβαίω και τα κράτη-μέλη, όπως είπα και προηγουμένως, και η αυτοκινητοβιομηχανία ε, και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συνεργαστούν όσο γίνεται περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ε, λύσεις στο, ε, σύστημα, στο πρόβλημα αυτό. Δεν θέλουμε να υπάρξουν ανώφελες ε, καθυστερήσεις σε όλα αυτά τα συστήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια των πολιτών. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την διαρκή στήριξη που παρέχετε στην ε, ανάπτυξη του, της υπηρεσίας e-call ε, και νομίζω ότι είναι σαφές ότι εάν ε, δουλεύουμε όλοι μαζί, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα από ότι αν ο καθένας δουλεύει από τη δικιά του την πλευρά. Και γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι προσπαθούμε να συνεργαστούμε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε όσο γίνεται γρηγορότερα να δώσουμε την υπηρεσία αυτή τους πολίτες μας. Αυτό θα είναι περίπου, ε, αυτός θα είναι ε, ο εξοπλισμός. Ε, σχεδόν μπορεί κανείς να το φορέσει και σαν καρφίτσα στο πέτο του. αστείευομαι βέβαια. Πάντως αυτό αυτό το πολύ μικρό πραγματάκι ε, μπορεί να παράσχει εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Βλέπω ε, ότι είστε ήδη εξοπλισμένοι. Θα δώσω το λόγο για σύντομες ερωτήσεις. Επιτρέπετε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κύριος Κόχ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ ωραία ακούγονται αυτά, κυρία Κρούς, όταν τα ακούει κανείς για πρώτη φορά. Εγώ πριν από 10 χρόνια ε, ε, έκανα την πρώτη μου εμπειρία. Κάλλας, Ταγιάννη, Δε Παλάσιο, Φερχόιγεν ε, και άλλοι και η κυρία Ρέντινγκ τα ίδια είπανε. Τα κράτη-μέλη όλα υπογράφουν το μνημόνιο κατανόησης, όχι μόνο 22 και τα 27 κράτη. Ε, δεν θα είναι μόνο για τα γιοταχή και για τα ελαφρά φορτηγά, αλλά και για τα βαριά φορτηγά, για τα ε, λεωφορεία και για τις μοτοσυκλέτες, όπως θα λέει η εκθεσή μου. Από το 2015 λέτε μπορεί να εφαρμοστεί. Εδώ και 10 χρόνια τα ακούω αυτά τα πράγματα. Συγκεκριμένους χρόνους θέλω ημερομηνίες. Γιατί υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις και ποιες είναι αυτές. Μας είπατε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Μια ζωή καθυστερήσεις ακούμε. Συγκεκριμένα πότε θα έρθει αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Ε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και ε, του εισηγητές. Χαίρομαι που σας βλέπω και εσά και το επιτελείο σας που αναπτύσσετε αυτή. Και πραγματικά ξέρω ότι είστε προσιλωμένοι σε αυτή τη προσπάθεια, αλλά δεν εξαρτάται 100% από εμά. Συμφωνώ ότι η εθελοντική προσέγγιση μέχρι τώρα δεν μας οδήγησε σε ικανοποιητικά επαρκή επάση περιπτώσει αποτελέσματα και χρειάζεται μελέτη αντικτύπου. Τα κανονιστικά μέτρα είναι τα καλύτερα, για να μην πω τα μόνα σωστά. Το τεχνικό ζήτημα είναι καθοριστικό. Οι εταιρείε ε, κινητής τηλεφωνίας ε, πώς ε, θα πιεστούν ή πώς θα κληθούν να υποστηρίξουν αυτό το σύστημα και πώς θα μπει σε όλα τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να μπει και στα FEE λεωφορεία και στα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Τα FEE όμως για είναι πιο ακριβά από τα κανονικά. Επίσης η Επίτροπος Κρούς λέει ότι δεν χρειάζονται μόνο κοινέ ε, ρυθμίσεις και τεχνικές προδιαγραφές αλλά και κοινή ε, υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός. Έχετε δίκιο. Ε, αλλά χρειάζεται και κάποια πίεση. Τι γίνεται με εκείνους που είναι ακόμα διστακτικοί και δεν υπογράφουν. Τι γίνεται με τους πολίτες. Πώς θα τα μάθουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάνετε καμιά διαφημιστική εκστρατεία. Και αν ναι, πότε προτίθεστε να τη λανσάρετε. Καταλήτης λέτε είναι, είναι καταλήτης αλλά είναι αποτελεσματικός, μπορεί να σώζει 5.000 ζωές. Όπως ε, ρώτησε κάποιος συνάδελφος ε, σε μια ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα όμως έχει σκαλώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τα στοιχεία τα ξέρουμε, τα ωφέλη τα ξέρουμε. Το επόμενο βήμα που θα κάνετε, ποιο θα είναι και πότε. Το συντομότερο ελπίζω. Και τι φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για το γεγονό ότι τα πολύ σοβαρά τροχιά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη γίνονται σε αστικέ και περιαστικέ περιοχέ. Και πάλι σα ευχαριστώ για τι προσπάθειέ σα και ε, πιστεύω ακράδαντα ότι η Επιτροπή μας θα κάνει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για να σας υποστηρίξει. Ευχαριστώ, Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Επίτροπο για την έκθεσή της. Βεβαίως, το είπατε, είναι τεράστια σημασία η έρευνα για μας και έχουμε τη δυνατότητα να σώζουμε ζωές. Πολλά θέματα ε, συζητήθηκαν από τους προλαλήσαντες και επίση καλό θα ήταν να μην μείνει αυτή η προσπάθεια γιοταθεί. Έχω όμω και άλλε ερωτήσει που δεν έγιναν ακόμα. Πρώτα είπατε, ο στόχο είναι μέχρι το 2015 να μπει σε όλα τα νέα γιοταχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ECOL, call Ε, και τα παλιά τι γίνεται, μπορεί να μπει αυτό ο εξοπλισμό έξτρα, το έχετε συζητήσει ήδη με του κατασκευαστέ. Ε, στη συνέχεια, τι γίνεται με τα οικονομικά. Υπάρχει και οικονομικό εμπόδιο ε, υποδομή και ένα τρίτο σε όλα τα συστήματα ενημέρωσης που έχουμε υπάρχει και ένα ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το Equal που είναι κλίση έκτακτης ανάγκης βεβαίως ε, προσφέρεται για λιγότερες ε, καταχρήσεις. Αν συνδυαστεί όμως με τα συστήματα πλοήγησης υπάρχει κίνδυνος. Ε, λοιπόν προστατεύονται τα δεδομένα και πώς το βλέπετε αυτό και πώς θα το παρακολουθείτε. Ευχαριστώ κύριε Μάισνε. Και κυρία Φώστερ. Thank you, Ευχαριστώ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, κοιτάξτε με, ναι. είναι δύσκολο να, πάρουμε, να έχουμε μια ορθολογική προσέγγιση απέναντι σε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και προκαλούν έτσι μεγάλη ε, ευαισθησία στον κόσμο. Εγώ πάντως θέλω να συμφωνήσω ε, με αυτά που είπε η κυρία Μάισνερ προηγουμένως εάν έχουμε ε, κάποια, ε, αν είχαμε σε εθελοντική βάση εφαρμογή αυτών των ε, προγραμμάτων, δεν θα είχαμε πρόβλημα κανένα και εγώ προσωπικά δεν θα είχα. Απ' την άλλη πλευρά, δεν ξέρουμε καθόλου ποιο είναι το κόστος για την αυτοκινητοβιομηχανία της ενσωμάτωσης του εξοπλισμού αυτού. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, φυσικά. Εάν θέλω να αγοράσω, ας πούμε, ε, να αγοράσω ένα αυτοκίνητο το 2015, αλλά δεν θέλω, δεν επιθυμώ να έχω τον εξοπλισμό αυτό ε, στο αυτοκίνητό μου, γιατί δεν θέλω να μπορεί να με ανοιχνεύσει οποιαδήποτε αρχή, οποιαδήποτε στιγμή ταξιδεύω με το αμάξι μου. Τι θα κάνω. Ε, επομένως, ε, ή, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να έχουμε δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Είναι λίγο να θέλουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Τι να σας πω. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη αλλά να μην ε, έχουν ε, τη διάθεση να μπορεί κανείς να, γνωρίζει οποιαδήποτε στιγμή που βρίσκονται. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό τον εξοπλισμό. Δεν είναι πολύ σαφές και δεν είναι τόσο απλό όσο μερικοί και τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φώστερ Κράμερ. Ναι, μπορώ να συνεχίσω. Ευχαριστώ για την αναφορά και την παρουσίαση, αλλά τα συζητάμε πολλές φορές και το θέμα της προστασίας των δεδομένων είναι αποφασιστικό και θα πρέπει να λυθεί όπως και το κόστος. Όχι μόνο το κόστο του αυτοκίνητου, αλλά η σύνολη υποδομή. Πόσο υψηλό είναι και ποιο το υπομίζεται. Και μπορώ να συνεχίσω. ε, αυτοκινητοβιομηχανία ήδη μπορεί να το παρέχει εθελοντικά και μπορεί ο καθένας να αποφασίζει. Ούτε στη Γερμανία σε όλα τα κρατήδια ακόμα δεν έχει εισαχθεί. Ε, ας πούμε να έχουμε ένα σύστημα ε, για περκαγιά στα νοικοκυριά, στα σπίτια. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολλά τροχέα με νεκρούς και τραυματίες που μπορούν να σώνονται με αυτό το σύστημα. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και πόσο είναι το κόστος και ποιος θα το πληρώνει. Όχι μόνο μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί χρειάζεται και υποδομή. Και ποια άλλα είναι τα υπόλοιπα μέτρα που δεν σκεφτόμαστε ε, να το εισαγάγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή πανευρωπαϊκό. Όποιο θέλει τέτοια προστασία αγοράζει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι υποχρεωτική αυτή η ε, συσκευή. Όποιο θέλει όμω μπορεί να την αγοράσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κράμε. Α, κάτι ξέχασα, συγγνώμη. Για παράδειγμα, ε, μου έστειλε επιστολή ο επόπτης ε, προσωπικών δεδομένων στη Γερμανία. Στα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα ρωτάει πώς θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Είναι μεγάλο πρόβλημα να μπορεί ο καθένας να σε παρακολουθεί, να ξέρεις που είσαι ανα πάσα στιγμή και που κινείσαι και που βρίσκεσαι. Ευχαριστώ η κυρία Κρούς για να απαντήσει στις ερωτήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζοντας θα σας επαναλάβω ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο αποφασίστηκε στο γόνατο. Ούτε είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τη δική μου υπηρεσία, τους συναδέλφους στην ε, Επιτροπή επίσης. Πρόκειται για από εκεί μας στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. και έτσι θα αποκτήσετε περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτή τη ρύθμιση και επίσης έτσι έχετε και κάποιες ε, εγγυήσεις για το ότι έχουν γίνει ιδέουσες ε, σταθμίσεις ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση. Πέραν αυτού. Εάν θεωρείτε ότι είμαι θα ότι πρόκειται να φτάσουμε εκεί ε, με το 2015 όσον αφορά τη ρύθμιση με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για του άλλου εμπλεκομένους. Είναι αυτό το σίγουρο. Εγώ είμαι σίγουρη. Και αυτό η μελέτη των επιπτώσεων ε, ανέθεσε αυτή την, ε, τη ρύθμιση στους ε, ιδιώτες, στον ειδικό τομέα, αλλά αυτό είπαμε ότι δεν αρκεί, διότι έχουν περάσει 10 χρόνια και παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, οπότε πάμε στο 0,5% του συνόλου των αυτοκινήτων το οποίο είναι εξοπλισμένο κατά τον τρόπο οπότε επομένως για να γίνει αυτή η παράλληλη εφαρμογή αυτό χρειάζεται δέσμες από όλους τους εμπλεκομένους και αυτό επίσης ε, ε, θα προχωρήσει σύμφωνα με την πρότασή μας την νομοθετική γνωρίζουμε ότι τα θέματα τα οποία απασχολούν κάποια κράτη-μέλη ε, είναι υπαρκτά, τα καλύψουμε και προχωρούμε σε συνεργασία με τι αρμόδιε υπηρεσίε, οπότε θεωρούμε ότι θα βρεθούν οι κατάλληλε λύσει, ώστε να προχωρήσουμε σε αυτήν την εφαρμογή τη ρύθμιση για το e-call. Ε, Επίση, θα υπάρχει μια σχετική εκστρατεία ενημέρωση για τον κόσμο και αυτό το προετοιμάζουμε και πάλι σε στενή συνεργασία με του εμπλεκομένου, γιατί αυτό θα γίνει του χρόνου. Και η ομάδα που ασχολείται με αυτό προσπαθεί να δει πώς θα καλυφθούν και τα οικολογικά αυτοκίνητα. Δεν το ξεχνούμε αυτό. Είπαμε επίση να δούμε ένα αυτοκίνητο πώ το κόστο θα συγκρατηθεί κάτω από τα 100 ευρώ. Και βεβαίω δεν θα σα εξηγήσω το πόσο μας απασχολεί το θέμα της προστασία των δεδομένων και εν προκειμένου και γενικότερα. Αυτό δεν θα σας εκπλήξει. Ξέρετε άλλωστε το παρελθόν μας. Μην ανησυχείτε. Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Και θεωρούμε ότι προτεραιότητα εδώ έχει η ασφάλεια. και ελπίζουμε ότι θα συντονιστείτε με τις προσπαθειές μας και αν κάποιος θέλει το 2015 ερώτα να αγοράσει ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να φροντίζει για το τι θα κάνει εάν πρόκειται να προβεί σε κάποια αντικατάσταση ή όχι και δεν ξέρω αν τι θέλετε να απογίνει με το αυτοκίνητο, αλλά τέλο πάντων δεν ξέρω τι εναλλακτικέ έχετε. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, το βαθμό, τόσο το, τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα βρει τη λύση του με το μέτρο αυτό. Επίσης, θέλω να σας αναφέρω και κάτι άλλο. Το θέμα του τι θα γίνει με το 2015 με αυτή τη ανακοίνωση και θέλω να σε εξηγήσω ότι εάν κανείς διαλέξει το αυτοκίνητο για να πάει στον προορισμό του θα πρέπει να λάβει υπόψη τους κανόνες που ισχύουν. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μεγίστη δυνατή ασφάλεια. Όποτε υπάρχει κάποιος κίνδυνος, να υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει κανείς βοήθεια. Τώρα, επανέρχομαι στο θέμα της προστασίας των δεδομένων νομίζω ότι έχει αντιμετωπιστεί ισορροπημένα το θέμα, γιατί από τη μία μεριά δεν θέλουμε να α, ε, κοινοποιείται το μέρος που βρίσκεται κανείς, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να εξασφαλιστεί ε, το ότι θα προστατευτεί η ζωή αυτών που κινδυνεύει, κάτι το οποίο έχει προτεραιότητα και για να γίνει αυτό θα πρέπει ε, να γνωστοποιηθεί ε, τοποθεσία που βρίσκεται. Και εδώ μιλάμε για κάποιο σοβαρό περιστατικό. Α, και κάτι άλλο, ίσως να σας ε, αναφέρω. Κάτι το οποίο το έχει προτείνει ο κύριος ε, Κράμερ ότι ενεργοποιείται η συσκευή μόνο όταν σταματήσει με τρόπο υποχρεωτικό, καταναγκαστικό, βίο, αν θέλετε, το ε, όχημα. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, νομίζω ότι δείξατε ότι είσαστε αποφασισμένοι τόσο ώστε να μπορέσετε να διεκπαιρεώσετε αυτό το, το, το, θέμα το οποίο εκκρεμούσε τόσο καιρό και και όλος ο κόσμος ελπίζει ότι το σύστημα αυτό θα μπορεί να τρέχει από το 2015. Υπάρχει δηλαδή και το δίκτυο θα μπορεί να τρέξει ακριβώς το σύστημα, κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. αυτά τα μέτρα, αυτές τις προτάσεις και σας ευχαριστούμε που μας τις ε, παρουσιάσατε. <clears throat> Euh, Συνεχίζουμε λοιπόν με την Επιτροπή. Καλωσορίζω τον κύριο Τιμπέκα που αντικαθιστά τον αγαπητό μας φίλο Ντίρκ Στέξ, ο οποίος μας παράτησε, σηκώθηκε και έφυγε. Θα ανακοινωθεί στην επόμενη Ολομέλεια ε, η σχετική δήλωση ε, για την ιδιότητά του ως νέο μέλος, ωστόσο έχει έρθει ο νέος συνάδελφος. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ως ήθιστε, θα παρακαλούσα πρώτα τους συναδέλφους να μας πούν ποιος έχει ξεχάσει την κάρτα του. ο Ματιέ Γκρός, καλά. Άλλος της... Μόνο ο Γρός. Εντάξει. Λοιπόν, με τις κάρτες ψηφίζουμε. Ε, να κάνουμε μια μικρή δοκιμή όπως συνηθίζουμε. Και θα σας παρακαλέσω να ψηφίσετε, σας παρακαλώ. Σε κοντέ. Ben, <laughs>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 Euh, euh, λοιπόν, πάμε στην κανονική ψηφοφορία τώρα. Euh, το θέμα είναι συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Πράσινο Ακροτηρίου. Εδώ μόνο ναι ή όχι μπορούμε να πούμε. Τροπολογίες δεν έχουμε. Εγώ είμαι ο εισηγητής. Απλώς, παρά το χαρακτήρα το σχετικά μικρό του Πράσινου Ακροτηρίου, η συμφωνία είναι πλαίσιο, ε, απεριόριστη και είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα αυτή, για τα νησιά του Πρασινού Ακροτηρίου, γιατί περίπου το 100% της οικονομίας τους εξαρτάται από τον τουρισμό και μέγα μέρος των τουριστών αυτών είναι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό και η συμφωνία με τα 27 κράτη-μέλη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα. Λοιπόν, απουσία τροπολογιών και δεν θέλει κανεί να μιλήσει, να πει τίποτα σημαντικό, Σα προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευρωπαϊκή Ένωση Πράσινο Κρατήριο. Α, θέλει η κυρία φώστε να μιλήσει. Όχι, η ΓΟΥΙΠ είναι και δεν είναι σήμα. Α, είστε ΓΟΥΙΠ, μάλιστα. Καλά. Καλώς. Δύο είστε. Άλλος. ε, ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζετε διανατάσσεω τη χειρό. Έχετε ξεχάσει και εσεί την κάρτα σα. Όχι, δίνει γραμμή. Πέρας. Ε, ψήφισαν 29, 28 υπέρ και ο κύριος Ματιό Γκρός χωρίς κάρτα. Σας ευχαριστώ και περνούμε στη δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία που είναι το μέλλον του ΦΠΑ, του φόρου θέμες αξίας. Μια στιγμή. Προσθέστε και τη δική μου ψήφο παρακαλώ. Νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή ψηφοφορία. Ψήφισα δυνατά στους χείρους. Είχα κάρτα από όλα, αλλά δεν κατάλαβα ότι ψηφίζαμε και ξέχασα να ψηφίσω ηλεκτρονικά. Ωραία. Ε, πάμε λοιπόν στο μέλλον του ΦΠΑ και θα παρακαλούσα τον κύριο Φέρμπερ να μας πει αν έχει να κάνει σχόλια για την έκθεσή του ή αν μπορούμε να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία, αν έχει τίποτα προσθέσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε μόνο συζήτηση πριν την κατάθεση τροπολογιών και δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Δέλφους που ε, και το καλοκαίρι έκαναν τροπολογίες, προσπάθησα όσο μπορούσα να λάβω υπόψη μου αυτά που ζητούν. Παρακαλώ μόνο την κατανόησή σας να καταλάβουμε ότι πρόκειται για το ΦΠΑ. Εμείς είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο ΦΠΑ των μεταφορών. Σε θέματα που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής πραγματικά και που χρειάζεται και δράση. Γνωρίζουμε κατά τα άλλα ότι υπάρχουν ε, ε, εδώ και χρόνια πολλές εμπλοκές για νομοθεσία για το ΦΠΑ, ας πούμε. Για το ταχυδρομείο, όλες Σμιτ που είχε διατελέσει, αν θυμάστε, ε, εισηγητής ε, για το ΦΠΑ στο ταχυδρομείο από τότε που τα ψηφίσαμε, που δεν θυμάμαι πότε ήταν ε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, έχει φρακάρει στο Συμβούλιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να προχωρήσει, αλλά τι να κάνουμε είναι δύσκολο γιατί ξεπερνά κατά πολύ τα όσα έχουν γραφτεί στο έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είμαι και μέλος στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων που είναι επί της ουσίας αρμόδια και νομίζω θα το συζητήσουμε και εκεί στην τελευταία έκθεση που θα καταθεί στην Ομέλεια, γιατί τούτη εδώ είναι γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φέρβερ. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε τότε. Έχουμε κάποιες τροπολογίες. Είστε έτοιμοι. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας σας όλοι με τη σειρά της τροπολογίας. Πάμε. Η τροπολογία υπαριθμών 1 είναι του εισηγητού. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά... Όχι, είναι του κυρίου Ρικέ. Η τροπολογία εισηγητής είναι υπέρ. Αποχές. Ευχαριστώ. Η τροπολογία υπαριθμών 2, εκράμερ ο εισηγητής αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τρία. Euh, εισηγητής κατά ψήφι υπέρ της τρία της κυρίας Τσικαού. Κατά. Απορρίφεται. Τσεκ. Καλά, θα το ελέγξουμε. Ε, ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 3. Ε, δεν ανοίγει η ψηφοφορία ο νούπο, τώρα λίγο θα ανοίξει. Τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Α, λοιπόν, Ποιο ψηφίζει χωρίς μηχάνημα υπέρ. ο χειρό. Κανείς. Κατά. Δύο. Άρα 17 κατά, 14 υπέρ, άρα απορρίπτεται η τροπολογία. Η τροπολογία που αριθμό 4. Κράμερ Ντυρό. Ο εισηγητή είναι κατά. Ψήφι υπέρ. κατά νομίζω ότι είχε απορριφθεί ε, τροπολογία παριθμό 5 κράμερ τυρό ο εισηγητή κατά ψήφιπε. κατά νομίζω ότι απορρίπτεται η έξι της κυρίας Τσικάου ο εισηγητής επίσης κατά ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται επίσης. Η επτά του κυρίου Τρεμόσα. Ο εισηγητής είναι κατά ψήφι υπέρ. Κατά. εποχές. Νομίζω ότι είχε απορριφθεί και αυτή η τροπολογία του κυρίου Ρικέ. Ο συγκεκριτής είναι αντίθετος. Ψήφι Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Οι τροπολογίες 9 και 11 μαζί, Βαντάλεν και Πάξας, γιατί είναι ταυτόσιμες. Ο εισηγητής είναι αντίθετος. Ψήφι πέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 9. Το δεύτερο τμήμα του κυρίου Βαντάλεν. Ο εισηγητής είναι κατά. Ψήφι Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παρθών 10. Κράμερ Ντουιρό. Ο εισηγητής είναι κατά. Ψήφι Πέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία του κυρίου Πάξας, το εισηγητής είναι αντίθετος. Ψήφι Πέρ. Είναι η 11. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 12. Στέρξ. Εντάξει, να είστε βιανικοί με τον συνάδελφο. Υπέρ. Και η υπέρ είναι. Κατά. Ορίστε. Ε, τιμητική έγκριση κατόπιν αποχωρήσεως του συναδέλφου. Ε, επόμενη, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Είναι συμβαστική α. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε κατά πίπτη 15 Κράμερ και Ντουιρό. Μάλλον. Διότι εγκρίθηκε προηγούμενα και πάλι στη 13. Το κύριο Μπαλτσίτη. Ο εισηγητής κατά ψήφι Κατά. Απορρίπτεται. 16. Έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά τμήματα. Α, συγγνώμη, ξέχασα τη 14, λέει ο πρόεδρο. Πρέπει να ψηφίσουμε. Του κυρίου Παξά. Ο εισηγητή είναι κατά. Ψήφι Κατά. Η τροπολογία αυτή απορρίπτεται. Η 16 τώρα του κυρίου Δανέλη έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία σε τμήματα. Το πρώτο μέχρι του στόχου, ο εισηγητή είναι υπέρ, ψήφι υπέρ, του στόχου ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των μεταφορών. Κατά. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο, μετά του στόχου. Ο εισηγητή είναι αντίθετο, ψήφι υπέρ. Ε, κατά. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Το 17 τώρα του κυρίου Ρανέλη είναι κατά ο συγκεκριτής, ποιοι είναι υπέρ. Qui vote contre. Ποιοι είναι κατά. Euh, je pense qu'on peut faire un check peut-être pour vérifier, mais je pense que cet amendement est repoussé. Νομίζω ότι απορρίπτεται, οπότε να κάνουμε όμως την ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Είκοσι, έντεκα. <coughs> Euh, Και τώρα πάμε στην παράγραφο 6. Υπάρχει μια συμβαστική πρόταση του συγητού, ποιοι είναι υπέρ του, της συμβαστικής διατάξεως Β, ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται, οπότε η τροπολογία 18, η 18 διορθώνει ο μιλητής, καταπίπτει, αλλά έχουμε τώρα να ψηφίσουμε την 19 του κυρίου Πάξα Πάξας ε, κατά ο συγκεκριτής, ποιοι είναι υπέρ του 19, ποιοι είναι κατά. Οπότε, απορρίπτεται. Υπαριθμόν 20 τώρα, Φαντάλεν. Κατά. Mm. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Να κάνουμε τώρα την λειτουργική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 18-17 και τώρα 21 ε, φιντάντζα είναι υπέρ ο συγκητής Ποιοι είναι υπέρ Ποιοι είναι κατά εγκρίνεται Έξι, νέα, Και εδώ υπάρχει πολύ σημαντική πρόταση του εισηγητού. Είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε και καταπίπτουν οι 22 και 23. Και τώρα κάνουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. 28, 3 και μια αποχή. Επομένως, θα πρέπει να συγχαρούμε τον εισηγητή. Οπότε θα πάει στην Ολομέλεια η συμφωνία για προς στο κρατήριο ε, για την Ολομέλεια του Οκτωβρίου και τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του ΦΠΑ. Έχουμε για εδώ πέρα ε, την, την έκθεση αυτή που θα συζητηθεί στις 19 ε, και πάμε τώρα στην Λευκή δουλειά για το μέλλον των μεταφορών και τον λόγο έχει ο εισηγητής ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μερικά εισαγωγικά σχόλια για την έκθεσή μου. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι αυτή είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας. Και μας δεσμεύει και ο αριθμό των σελίδων, τέσσερις συγκεκριμένα. Ε, κανονικά θα θέλαμε να γράψουμε πολλά περισσότερα, χωρίς να το διακινδυνεύσουμε για το μέλλον να γίνει τόσο μεγάλη γνωμοδότηση που να μην έχει κέντρο βάρους και ε, ουσία. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις πολιτικές ε, ομάδες για να επεκταθεί η γνωμοδότηση, αλλά παραμένει η επιθυμία μου να είναι σε ένα λελογισμένο πλαίσιο ε, και έτσι κάπως συμπυκνωμένη η γνωμοδότησή μας για να έχει και ουσία. Αυτό Επίσης σημαίνει ότι ό,τι δεν έχω συμπεριλάβει δεν σημαίνει ότι είμαι απαραίτητος αντίθετος ούτε απαραίτητος υπέρ. Οπότε μην κάνουμε τέτοια συζήτηση. Ε, είναι δεδομένη η έκταση. Τι να κάνουμε. Κάτι άλλο. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα το 2010 και στην Επιτροπή μας και στο ε, Κοινοβούλιο συνολικά για το μέλλον των μεταφορών. Εγώ είχα το καθήκον βεβαίως να δείξω μια συνέπεια και με τις βασικές αρχές ε, της έκθεσης αυτής και στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτό. Γιατί έτσι θα είμαστε και πιο πιστικοί και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέναντι και στο Συμβούλιο. Λευκή βίβλος λοιπόν για περίοδο μέχρι το 2050. Το προεξοφλώ από τώρα. Για μένα ήταν σημαντικό βεβαίως ε, να μην χάσουμε το στόχο του 2050 και σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ και με το στόχο του 2050, αλλά είναι και προς το συμφέρον της συγκεκριμένης πολιτικής, του στόχους μας να τους προσανατολίζουμε και να τους ορίζουμε για πιο σύντομη περίοδο Γι' αυτό πρότεινα 2010-2020 ε, ε, και να τολμήσουμε και ένα βλέμμα προς το παρελθόν, γιατί και το 2010 κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον των μεταφορών. Για να δούμε ε, ποιους στόχους καταφέραμε να πετύχουμε του 10, ε, ποιους δεν πετύχαμε και πώς τα εφαρμόζουμε. Έχω βάλει δύο παραδείγματα πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου. Το ένα που αφορά τη ε, οδική κυκλοφορία και το θέμα της ασφάλειας δεν έχουμε πετύχει όλους τους στόχους μας, αλλά κάτι που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είχαμε βάλει ένα στόχο με αριθμητικά στοιχεία και κάθε χώρα ε, αισθάνθηκε υποχρεωμένη να ε, καλύψει αυτό το ποσοτικό στόχο. Και τελικά είχαμε επιτυχία. Αντίστοιχο λοιπόν πρόγραμμα θα μπορούσαμε να προτείνουμε για τα έτη 10-20. Κάτι άλλο αρνητικό ως εμπειρία ήταν η εσωτερήκευση του κόστους. Αυτό που καταφέρουμε στην οδική κυκλοφορία είναι ένα μέρος των όσων περιμέναμε μόνο και είναι καλό παράδειγμα αυτό που πρέπει να επανεξετάσουμε και προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα τελευταίο πάλι ως προς την ανασκόπηση είναι η εφαρμογή των όσων αποφασίσαμε θα το πω έτσι λίγο απλά, αλλά στα ράτα. Εκπλήσωμαι κάπως που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πιο επικριτική σε αυτό το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίησης, παρόλο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι από τα μεγαλύτερα αγκάθια του παρελθόντος. Θα το πω έτσι, ως εξής. Όταν είναι καλή η εφαρμογή, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, οι στόχοι του 2000 να εφαρμοστούν. Αν είχαν γίνει όλα αυτά, σήμερα θα ήταν η υποδομή καλύτερη και οι μεταφορές θα ήταν καλύτερες στην παροχή υπηρεσιών, ε, ακόμα και στις συνθήκες απασχόλησης, βλέπε μισθή, και θα είχαμε και καλύτερη κατανομή των μεταφορών στους διάφορους τρόπους και μέσα. Αν ήταν αυτοί οι στόχοι μας και παραμένουν, ε, λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε το Συμβούλιο και να πούμε ειλικρινώς ότι δεν έγιναν κάποια πράγματα και να ρωτήσουμε γιατί δεν ε, ε, επενδύουν σε κάποια μέσα μεταφοράς για να είναι αύριο πιο ελκυστικά. Αυτό θέλω να ε, μπει στην έκθεσή μου, να παραμείνει και να αποδώσουμε και τις ευθύνε εκεί που ανήκουν. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε τους καλύτερους νόμους και να συζητάμε και έχουμε συζητήσει και για το σιδηρόδρομο, είχαμε συζητήσει και για το ΕΡΙΚΑ. Ε, το κοινοβούλιο δεν είναι παράλογο, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση να εφαρμοστούν αυτά. Γιατί σε πολλά κράτη υπάρχει ακόμα εντύπωση και η πεποίθηση ότι με οικονομικό προστατευτισμό υπηρετούν τις μεταφορές, ενώ είναι εντελώς το αντίθετο. Αυτά, εισαγωγικά. Γενικά πάντως θα έλεγα ότι οι στόχοι μας συνδέονται πάρα πολύ με αυτά που είχαμε συζητήσει το 2000 θα πρέπει τα διάφορα στοιχεία και τις εξελίξεις να τα επικαιροποιήσουμε και ο στόχος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενέργεια, για την κινητικότητα ε, γενικά, για την κατανομή στις, ε, στα διάφορα μέσα μεταφορών παραμένουν. Αν θέλουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, δύο είναι οι δρόμοι το ένα είναι να καταργήσουμε τα εμπόδια που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει ως ενιαίος χώρος. Εγώ μ' αρέσει να μιλάω για ε, τις επιπτώσεις ε, τις συνοριακές ε, και στην τεχνολογία και στην νομοθεσία και στην πράξη. Αυτά είναι εμπόδια στις παραμεθόριες περιοχές. Εκεί μπορούν να ληφθούν μέτρα πάρα πολύ γρήγορα στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας, το έχω ξαναπεί, και στην αιτιολογική έκθεση. Αν γνωρίζουμε σήμερα ότι έχουμε 6.000 ρυθμίσεις, 6.000 κανόνες για το σιδηρόδρομο που δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκό συνδρόμος και από τις 6.000 κανόνες περιτεύουν οι 4. Γιατί δεν μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι ε, τον ευρωπαϊκό χώρο χωρίς να ξοδέψουμε ούτε δεκάρα. Απλώς πολιτική βούληση χρειάζεται και πιο ευρωπαϊκή αντίληψη. Είναι καλό παραδείγμα ο σιδηρόδρομος, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και έχω βάλει και ημερομηνία. Νομίζω ότι έγινε καλή δουλειά στον οργανισμό θα πρέπει όμως να έχετε και τη δυνατότητα λήψης απόφασης για εφαρμογή σε όλων αυτών. Και αυτό θα ήταν καλό παράδειγμα, ότι ό,τι ζητάει το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να σκοντάφτει πάντα στα χρήματα. Ορισμένα πράγματα ε, σκοντάφτουν στην έλλειψη πολιτικής βούλησης. Βεβαίως χρειαζόμαστε και ε, να ανοίξουν οι αγορές. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Ε, για μας βεβαίως είναι αυτός ο δρόμος και αυτό το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη, αλλά η διάνοιξη των αγορών δεν θα πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε τίμημα και πάση θυσία. Υπάρχουν στοιχεία κοινωνικά, οικονομικά, οικολογικά και είναι όλα αυτά σημαντικά. Ένα άλλο στοιχείο στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου είναι και παραμένει το, τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν ξέρω ποια νέα ονομασία. Εδώ και 10, 15, 20 χρόνια ε, προσπαθούμε να σκαρφιστούμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα πολιτικό σθένος, να μειώσουμε τις προτεραιότητές μας, να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση και πραγματικά να βελτιώσουμε την κατανομή ε, αναμέσω μεταφοράς. Αυτό σημαίνει όμως ότι και χρονικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περίφημα bottlenecks, εκεί που έχουμε δυσκολίες τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και πάλι τα προβλήματα είναι στα σύνορα. Έχουμε διαπιστώσει ότι ιδιαίτερα στα σύνορα μειώνονται οι επενδύσεις γιατί δεν ενδιαφέρεται καμία χώρα από μόνη της να επενδύσει σε παραμεθόρια περιοχή αλλά από κοινού οι χώρες ναι. Και με τα διευρωπαϊκά δικτύα συνδέουμε και τη χρηματοδότηση. Δεν μου αρέσει αυτή η ιστορία του Ταμείου για τις μεταφορές, γιατί διαφώνησαν Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι νόμιζαν ότι ε, αυτό είναι ληστρικό. Δεν ξέρω πώς θα το πούμε, αλλά να το συζητήσουμε με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και την, Επιτροπή συγγνώμη, που είναι αρμόδια για την ενέργεια, για να βρούμε περισσότερους πόρους για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. και με νέα χρηματοδοτικά μέσα, με προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για να υπάρχει έτσι μια δυνατότητα ενίσχυσης ε, κάποιων ποσών που γράφονται ήδη στα άρθρα. Αυτά μπορούν να γίνουν συγκεκριμένα για το μέλλον. Αλλά θα πρέπει επίση να πούμε ότι δεν νοείται μια χώρα να χαρακτηρίζει ένα σχέδιο, ένα έργο προτεραιότητας επί 20 χρόνια. Ε, τι προτεραιότητα. Να φύγουν τα έργα που δεν αναπτύσσονται 20 χρόνια, γιατί δεν υπάρχει προτεραιότητα, δεν υπάρχει βούληση να προωθηθούν. Για την κινητικότητα τώρα και ιδιαίτερα για τις οδικές μεταφορές. Έχει πάρα πολύ σημαντική πτυχή εδώ η αστική διάσταση. Το 80% των πολιτών μας ζουν σε πόλεις ή στο μέλλον θα ζουν σε πόλεις. Εάν αυτό το θέμα το αφήνουμε στην επικουρικότητα και το ε, διεκπεραιώνουμε, έτσι λέμε δεν είναι δική μας υπόθεση, ξεχνάμε το 80% του πληθυσμού. Γι' αυτό προτείνω κι εγώ, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αστικές μεταφορές και η αστική ανάπτυξη να μας απασχολήσει περισσότερο. Οι αστικές μεταφορές θα πρέπει να είναι ε, συνδυασμένες με διάφορα μέσα μεταφοράς. Προσωπικά θεωρώ ότι στην οδική κυκλοφορία θα πρέπει να έχουμε ε, τις συγκοινωνίες, τις μαζικές, τις δημόσιες συγκοινωνίες, δημόσια με την έννοια της ε, παροχής υπηρεσίας, Ένα λεωφορείο μπορεί να αντικαταστήσει μέχρι και 50 αυτοκίνητα που είναι ο καθένας μόνος του. Αν είχα πάρει το λεωφορείο θα είχα έρθει μισή ώρα νωρίτερα που είχα φρακάρει το πρωί στο ποτηλιάρισμα. Λοιπόν, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, αυτά τα ζητήματα, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και κάνω μια γέφυρα τώρα ε, σε μια άλλη υπόθεση που θέλουμε να προχωρήσει και το συζητήσαμε το 2010. Όσο προχωράει καιρό χρειάζεται καλύτερη και σωστή κατανομή στα διάφορα μέσα των μεταφορών. Αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι δια αποφάσεων, να βγάζεις ένα φυρμάνι. Θα πρέπει και πάλι να ανταποκρίνονται, να είναι ε, αποδοτικές αυτές ε, οι μεταφορές, να λαμβάνουν υπόψη και την οικονομία και το περιβάλλον και την ασφάλεια των ενεχομένων ενεργητικά ή παθητικά και επίσης ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις συνθήκες εργασίας. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Αλλά ας μην τα υποτιμούμε αυτά τα θέματα γιατί αλλιώς θα παραμείνει στη θεωρία αυτό και να ξαναμπώ στα 300 χιλιόμετρα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με διάφορες προτάσεις 300 χιλιόμετρα, αλλά με ενισχύει το εξής. Σε ορισμένες περιφέρειες θα υπάρχει πολύ καλύτερη κατανομή κάτω από τα 300 χιλιόμετρα, σε άλλες περιφέρειες δεν θα υπάρξει ποτέ. είναι ευθύνη των κρατών και των περιφερειών να ορίσουν σήμερα στόχους και να μην τα ρίχνουν ο ένας τον άλλον για τη χρηματοδότηση και για τον προγραμματισμό. Ας μην κάνουμε τώρα δογματική συζήτηση και παίζουμε την κολοκυθιά 300 χιλιόμετρα. Υπάρχει και ένα άλλο μειονέκτημα στα 300 χιλιόμετρα και παραέρχομαι στην οδική ασφάλεια. Ε, ε, Πέρα από το συνολικό στόχο, κοιτάξαμε και τους στόχους που πέτυχε κάθε χώρα, που ήθελε ε, κάθε χώρα να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και να μειώσει τα θύματα από τροχέα, τους ε, νεκρούς και τους τραυματίες. Λοιπόν, χρειάζεται καλύτερη συνεργασία με τα κράτη γιατί ξέρουμε ότι κάθε χώρα κοινά από διαφορετική αφετηρία και ως προς την κατάσταση που επικρατεί και ως προς τις υποδομές. Και για τη φορολόγηση, δύο λόγια. Για μένα είναι πάντα ε, τα κίνητρα πιο ελκυστικά από ό,τι οι φόροι. Γιατί ο φόρος είναι συχνά διπλή και τριπλή φορολόγηση, γεμίζει μεν τα ταμεία, αλλά η συζήτηση για το earmarking και την εσωτερήκευση του κόστους μας έδειξε ότι όσο καλή πρόθεση και αν έχουμε, δεν βελτιώνει τη χρηματοδότηση των έργων. Ούτε εις δίτ, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υποδομές, υπάρχουν χρήματα, μπορούν να επενδυθούν στις υποδομές και θα επιφέρουν και έσοδα. Ε, αυτό δεν πέτυχε εν μέρη. Λοιπόν, για μένα αύριο το θέμα των τελών και των φόρων μπορεί να είναι ενδιαφέρον, διότι γεμίζουν τα ταμεία. Αλλά σας παρακαλώ, ας είμαστε προσεκτικοί. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά το θέμα που μας ενδιαφέρει εμάς δεν είναι να γεμίζουν ε, τα ταμεία τους Υπουργοί Οικονομικών και να αδειάζουν Υπουργοί Μεταφορών. Τελευταίο. Θα ήταν ενδιαφέρον εάν βλέπαμε εδώ τους στόχους. Έχω βάλει μια εικοσαριά στόχους, πολύ φιλόδοξους, το ξέρω. Δίνω τη δυνατότητα όμως και στην Κομισιόν να δείξει στο Συμβούλιο τι πίεση ασκούμε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και εκείνη πεπισμένη ότι είμαστε σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια και απέναντι μας έχουμε το Συμβούλιο. Αλλά είναι προς το συμφέρον και των πολιτών και της οικονομίας και του περιβάλλοντος να υπάρχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ένα αυτό. Δεύτερο. Διεθνώς μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι και να δείξουμε το δρόμο και στην έρευνα αν αρχίσουμε από σήμερα. Αλλιώς ε, αύριο θα μας έρχονται έξωθεν οι προδιαγραφές και μας τις επιβάλλουν, ενώ η Ευρώπη μπορεί να δώσει το παράδειγμα. Λοιπόν, σε αυτά τα θέματα χρειάζεται στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να χαθούμε στις λεπτομέρειες, να αναλωνόμαστε, να στείλουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο και μετά να μετράμε τους στόχους αυτούς. Κάθε 15 χρόνια, 20, 30, για να μην πω και κάθε χρόνο. Γιατί αν μετράμε τους στόχους κάθε πενταετία ή κάθε δεκαετία, Συχνά σκέφτεται ο σημερινό υπουργό ότι εντάξει μετά από μια πενταετία δεν θα είμαι εγώ, θα είναι άλλος. Είναι θέμα πολιτικής ευθύνης και για μένα παραμένει ζήτημα κλειδί η κινητικότητα. Γιατί αφορά όλους τους ανθρώπους, όλων των ηλικιών και καλό θα ήταν αυτούς τους στόχους να τους ε, τρούμε σε αιτήσια βάση, να τα δημοσιεύουμε και να λέμε τι πταίει. Ε, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ε, για τις τοποθετήσεις σας. Βεβαίως θα συνεργαστούμε με τις μεγάλες πολιτικές ομάδες όπως ήθιστε και με τις άλλες όπως ήθιστε σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Και εγώ δεν ενδιαφέρομαι να περάσω τις δικές μου ιδέες, πάση θυσία και να παλέψω με νύχια και με δόντια. Απλώς θέλω να μην ε, αναλωθούμε σε λεπτομέρειες, να μην χαθούμε και να έχουμε ένα σαφές μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, ματιού θα δώσω το λόγο στο σκιώδη συγητή να μην ξεπεράσει παρακαλώ τα τέσσερα, τους να μην ξεπεράσουν παρακαλώ τα τέσσερα λεπτά. Τέσσερα λεπτά λοιπόν για τους σκιώδης και ε, δύο λεπτά όλοι οι υπόλοιποι που θα πάρουν το λόγο γιατί διαφορετικά θα ξεφύγουμε τελείως ε, από τον χρόνο μας. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γκρός για την έκθεσή του είναι γεγονός ότι τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά τα θέματα και χαίρομαι που πολλά από τα όσα ζητήσαμε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο εκθεσής. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συστηματική του προσέγγιση, πώς ασχολείται με τα διάφορα μέσα μεταφορών και ε, τον ενδιαφέρει να είναι ε, σωστές οι συνδυασμένες μεταφορές και η διαλειτουργικότητα. Ωραία, συμφωνώ σε όλα αυτά. Αλλά εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και την αηφορία του όλου συστήματος. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον εισηγητή ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι μέχρι το 2020. Με μελέτες ε, και με ε, πραγματικά στοιχεία. Και μετά για τους στόχους που έχει θέσει μπορεί να είναι φιλόδοξη, αλλά θα πρέπει να είναι και ρεαλιστική. Ελπίζω να τα ξανασυστήσουμε αυτά τα θέματα αργότερα. Και θέλω να πω ότι στα συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να εξετάσουμε και τις μέχρι τώρα εξελίξεις. Σήμερα η κατάσταση διαφέρει το 2001 είχαμε ορίσει κάποιους στόχους σε μια λευκή βίβλο. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά ταυτόχρονα να κάνω και μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον καθορισμό των στόχων θα πρέπει να κάνει μια βαθιά ανάλυση της σημερινής κατάστασης και των υποδομών και ε, της ποιότητας των υπηρεσιών, της πυκνότητας του δικτύου. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες και παραμετρικοί. Επίσης έχουμε και νέες προκλήσεις Ιδιαίτερα η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Η ασφάλεια και η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστου σε όλα τα μέσα μεταφοράς είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνη. Επίσης, και οι αλλαγές στην οτροπία και στις συνθήκες και στις συνήθειες μετακίνησης του πληθυσμού θα πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι ο τρόπος που μετακινείται ε, πειράζει και το κλίμα και την ενέργεια και την κατανάλωση πόρων. Ε, θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, δημόσιες συγκοινωνίες στις αστικές και περιαστικές περιοχές. Θα βοηθήσει αυτό και το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική συνοχή. Επίσης, στις αστικές συγκοινωνίες Ε, βλέπουμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της ε, ε, οικονομικής κρίσης και των οικονομιών που πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη στους προϋπολογισμούς τους. Ξέρω ότι η οδική ασφάλεια είναι πολύ σημαντική στους αυτοκινητοδρόμους, αλλά το 70% των ατυχημάτων των τροχαίων γίνονται σε μικρούς δρόμους κακής ε, και όχι σε μεγάλου αυτοκινητοδρόμους. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα ε, διασυνοριακά έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν ε, εργαλεία της πολιτικής συνοχής και μέσα που μπορούν να βοηθήσουν και στην υπέρβαση των εμποδίων και των διαφορών που παραμένουν ακόμα ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Οι συνθήκες των εργαζομένων ε, είναι κάτι που μα ενδιαφέρει. Ε, μα ενδιαφέρει να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, η ασφάλεια των μεταφορών και η κατάρτιση των εργαζομένων. Επειδή όμως απελευθερώνονται οι υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ αυτό, τις συνθήκες ε, εργασίας. Ο εισηγητής Αναφέρθηκε στην αρχή των 300 χιλιόμετρων. Είναι στην παράγραφο 4 αυτό. Και λέτε ε, ότι θα πρέπει ε, να το δουν τα κράτη και οι περιφέρειες αυτό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια κεντρική ε, θεώρηση και ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και στην παράγραφο 6 αναφέρεστε στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές μέχρι το 2015. Μα θυμάστε τα προηγούμενα πακέτα και το πρώτο και το δεύτερο δεν πέρασε γιατί το ΕΛΚ αντιστάχθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνετε εκεί. κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ πολύ και εγώ και το Ματιό Γκρό και όλους τους ηγητές. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολη ήταν αυτή η προσπάθεια γιατί δεν έχει πολύ χώρο αυτή η έκθεση, δεν επιτρέπεται να επεκταθεί και το θέμα είναι πάρα πολύ ευρύ. Ήδη έχουμε συζητήσει αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές πρόκειται πραγματικά για το μελλοντικό προσανατολισμό των μεταφορών στην Ευρώπη με όλα τα στοιχεία και τις πτυχές που ανήκουν εκεί. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ε, ο Ματιό Γκρός και η Όλγα Σινιάλοβα γιατί ε, φαντάζομαι ότι θα τα ξέρετε κι εσείς και θα τα αναφέρετε κι εσείς. Γενικά χωρίς μεταφορές δεν μπορεί να λειτουργήσει η ενιαία αγορά. Και οι μεταφορές και η κινητικότητα είναι προϋπόθεση για αυτά που τάζουμε στην Ευρώπη, που υποσχόμαστε ελεύθερη κυκλοφορία, ελεύθερη ε, διακίνηση και μετακίνηση και για τους ανθρώπους και για τα εμπορεύματα και για τις υπηρεσίες. Ε, και θέματα ασφαλείας θέλουμε λιγότερους νεκρούς στους δρόμους ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα στο σιδηρόδρομο όπου δεν είναι συμβατά μεταξύ του για τεχνικούς λόγου, τα συστήματα, οι ράγες. Ή... Ε, στα ποτάμια έχουμε προβλήματα ακόμα στις εσωτερικές πλωτές ε, ε, οδούς. Τα δικαιώματα των επιβατών δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες ακόμα και θέματα κατάρτισης και πρόσβασης για μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι τεράστιο και ε, το πακέτο, εγώ μόνο εισαγωγικά ε, τα λέω αυτά και μπαίνω τώρα σε επιμέρους θέματα. Χαίρομαι που μιλάτε για συνδυασμό όλων των μέσων μεταφοράς. Το είδαμε όταν γνωρίσαμε την κρίση της ηφαιστειακής τέφρας, χρειάστηκε αλλαγή, εγκαταλείψαμε το αεροπλάνο και πήγαμε σε άλλους τρόπους και μέσα μεταφοράς και το όριο των 300 χιλιόμετρων που ανέφερε και ο κύριος Γκρος και η Όλγα συμφωνώ με τον εισηγητή χρειάζεται μια λύση πιο ευέλικτη όχι δηλαδή από τα 300 χιλιόμετρα και πάνω ποτάμια και σιδηρόδρομοι. Ποτάμια μπορείς να χρησιμοποιήσεις και σε λιγότερα από 300 χιλιόμετρα για λόγους οικολογικούς. Ή επίσης και πάνω από 300 χιλιόμετρα δεν είναι απόλυτο αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να διατηρηθεί ο αυτοκινητόδρομος όταν ε, δεν έχει σιδηροδρομικό δίκτυο ή δεν εξυπηρετεί, εν πάση περιπτώσει. Εγώ ζητώ λύσεις ευέλικτε από πλευρά τη ομάδα μου για περισσότερη ασφάλεια, φιλικότητα προς το περιβάλλον και αποτελεσματικότητα. Και ένα τελευταίο, τα εξής δύο, που είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο, και, και τα δύο αναφέρονται στην παράγραφο 16, στις πλωτές μεταφορές. Συμφωνώ με την Όλγα Σινιάδευα για το 2014 να έρθει μια πρόταση για τη ρύθμιση των λιμενικών υπηρεσιών. Γιατί χρειάζεται να αλλάξει τίποτα εκεί. Ήταν αρκετά δύσκολο το άλλο πακέτο για τα λιμάνια. Και τώρα θέλουμε πρόταση μέχρι το 2014 για τις λιμενικές υπηρεσίες με νέα μορφή. Γιατί αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ φιλόδοξο όσο και περιττό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε τι χρειάζεται και να γίνει. Και ένα δεύτερο, πάντα για τη 16, κάτι που μου λείπει εδώ, που είμαι και από το Βορρά, δεν θα πρέπει να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα στις εκπομπές, αλλά και το θείο. Με την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, η Βόρεια Θάλασσα και οι Βόρειες Θάλασσες γενικά έχουν άλλα διαφορετικά προβλήματα από τη Μεσόγειο. Να κοιτάξουμε το περιβάλλον παντού, γιατί οι εκπομπές θείου ε, βλάπτουν παντού και θα πρέπει σιγά σιγά να μειώνουν όχι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτά προς το παρόν εισαγωγικά και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ κυρία Μεσνέρ, ο Μάικλ Κράμερ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή, ιδιαίτερα για αυτό που μα είπε ότι δεν θέλει να επιβάλλει τι θέσεις του, αλλά να ζητήσουμε μια κοινή θέση απέναντι στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κυρίως απέναντι στο Συμβούλιο, γιατί ε, πρέπει να πετύχουμε και τους στόχους που έχουμε ορίσει. Οι μεταφορές οφείλονται για το 30% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ε, αυτό ε, είναι ήδη ε, πολύ σημαντικό. Αυξήθηκε πρόσφατα 35%, ενώ σε άλλους τομείς έχει μειωθεί ε, στα νοικοκυριά και στη βιομηχανία. Όλα τα στοιχεία και τα προβλήματα στις λευκές βίβλους που οφείλονται δεν κάναμε αναλύσεις στο τι φταίει. Κάνουμε ωραία κηρύγματα, ε, εξαγγελίες, μεγαλόστομα λόγια, προθέσεις, όλα αυτά είναι ωραία, αλλά γιατί δεν τα πετυχαίνουμε. Γιατί είναι πολύ χαμηλή η φιλοδοξία μας πρώτον στους στόχους. Η Κομισιόν είπε μέχρι το 2030 να μειωθούν και από το 2030 και μετά βλέπουμε ε, κατά 1% το χρόνο και μετά 5%. Αυτά είναι τώρα μπακάλικη λογιστική. Τι είναι αυτά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη μείωση από τώρα, αλλιώ δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουμε του στόχου. Παραπέμπουν τα προβλήματα στι καλένδε. Το μόνο που πρέπει να πούμε είναι μέχρι το 2020 στόχο τη Ένωση είναι μείωση κατά 20% και στι μεταφορέ τουλάχιστον 20% σε σχέση με το 1990. Αυτό είναι στόχο, όχι ένα ποσοστάκι το χρόνο. Αυτό λείπει από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δυστυχώς ματιού και από τη δική σου. Για να ξέρουμε πού θα μπει το ψαλίδι. Και ε, ο θέμητος ανταγωνισμός ε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπες ότι είναι καλύτερα τα κίνητρα από τη φορολόγηση. Αλλά τα καλύτερα κίνητρα 30 δισεκατομμύρια το χρόνο στην Ευρώπη, 30 δισεκατομμύρια δίνουν σε αεροπορικές εταιρείες. Μπορεί κανείς να πάει με μια τιμή ταξί από τη μια πρωτεύουσα στην άλλη. Ένα φοιτητή από το Βερολίνο που θέλει να πάει στο Παρίσι, ξέρω εγώ, το να πάει το αεροπλάνο γιατί είναι τόσο φτηνό. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε τι τάζουμε, τι υποσχόμαστε και είναι τρελό να τα πληρώνει πάντα ο σιδηρόδρομος. Κάθε μηχανή πληρώνει ένα τέλος στο σιδηρόδρομο, ένα διόδιο ας πούμε, και από, από 12 τόνους και πάνω τα φορτηγά στους αυτοκινητοδρόμους. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εδώ για φορολογία. Είναι το απλούστερο κίνητρο και το πιο φθηνό μέσο το αεροπλάνο. Δεν γίνεται αυτό. Μετά, τα μεγάλα έργα. Το τρίτο. Γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι ορισμένα μεγάλα έργα δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Ή σε 30, 40, 50 χρόνια. Βερόνα Μπολόνια η Ιταλία χρειάστηκε 80 χρόνια για να φτιάξει δεύτερη γραμμή. Και εσείς περιμένετε τα τρία μεγάλα ε, έργα να γίνουν. Ε, η σύραγγα Λιών το Ρίνο, ε, η σύραγγα στο Πολσάν, η γέφυρα στη Μεσίνη, στη Σικελία. Ποτέ τον ποτόν. Αλλά δεν τολμάει κανείς να πει να τα διαγράψουμε αυτά. Δυόμιση ώρες ε, πέρσι χρειαζόταν Βερολίνο Μπρέσλαο ε, ε, το τρένο. Σήμερα χρειάζεται 6 ώρες. Λείπουν 50 χιλιόμετρα ελάχιστα χιλιόμετρα μάλιστα για την ηλεκτροδότηση, αλλά για αυτά δεν έχει λεφτά η Deutsche Bahn, η γερμανική σιδηρόδρομη, αλλά πάνε και φτιάχνουν το σταθμό στη Στουτγάρδη, το Στουτγάρδη 21, το, το σούπερ έργο και η Πολωνία λέει 1,2 δις ε, για την αλλαγή ε, του τρόπου μεταφοράς. Είναι τρελά αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν χρήματα, αλλά τα δίνουν λάθο. Πρέπει οι προτεραιότητε να οριστούν διαφορετικά. σω να αυξηθεί και η συγχρηματοδότηση και η συνυπευθυνότητα. Δεν θέλουμε περισσότερα χρήματα στι μεταφορέ. Διαφορετική πολιτική χρειαζόμαστε. Λεφτά έχουμε. Μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα αν τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Και τα οικονομικά σε ένα σημείο γίνεσαι συγκεκριμένο 10% στι εσωτερικέ πλωτέ μεταφορέ. Εγώ έχω κατέβει το Δούναβι 100 χιλιόμετρα τη μέρα και συνάντησα τρία πλοία. Όλοι λένε για το Δούναβι. Μα δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχει ποτηλιάρισμα Δούναβη. Γι' αυτό αποφασίσαμε στο Κοινοβούλιο το 40% να πάει στο σιδηρόδρομο. 60% πηγαίνουν στον αυτοκινητόδρομο και 20 αυτή τη στιγμή στο σιδηρόδρομο. Εμείς αποφασίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία, το Συμβούλιο τα έχει στελώσει, για να το πω έτσι. 10% για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Δεν με ενδιαφέρουν εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο σιδηρόδρομος. Γιατί δεν βάζουμε εκεί όρια. Και λύγει και το θέμα της επιχωρικότητας. Βεβαίως θα πρέπει να λυθεί και το ζήτημα των πόλεων, αλλά δεν λύνεται έτσι. Δεν προχωρούμε και με τη χρηματοδότηση. Αλλά όσο δίνουμε 60% ε, ε, της πόλης στον αυτοκινητόδρομο, το θέμα δεν είναι να δίνουμε τα λεφτάκια σπάνω που θέλουν. Ε. Χρειάζονται πιο αυστηρά μέτρα και αυτό είναι δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς βέβαια να υπαγορεύει στις πόλεις τι πρέπει να κάνουν, να μην τα πετάμε από το παράθυρο. Μετά δεν θα μας εκπλήσουν, δεν χρειάζεται να μας εκπλήσουν τα κακά αποτελέσματα με απειλή ήδη ο πρόεδρος. Ε, περιορισμός ε, στην τα πανευρωπαϊκά. Ξέρουμε ότι στη Γερμανία 3% ε, θα έχουμε εξοικονόμηση και 30% μακροπρόθεσμα. Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που δεν έχει όρια ταχύτητας. Αν συνέβαινε παντού στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε περισσότερο θάρρος. Το ξέρω ότι δεν τα καταφέρνουμε αλλά και στην έκθεση ΚΟΧ είπαμε 30 χιλιόμετρα στις κατοικημένες περιοχές, ωραία, βεβαίως με τη δυνατότητα να υπάρχει κάποια ευελιξία. Ε, η Ευρώπη ε, δεν μπορεί παρά να βάλει το πλαίσιο στις προϋποθέσεις αυτές. Τα υπόλοιπα πρέπει να γίνουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτά. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε κοινέ λύσεις. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Επιτροπής των Περιφερειών. Παρακαλώ, είναι μεγάλη τιμή που σε έχουμε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τα μέλη της Επιτροπής σας που ε, μου απίθυναν την πρόσκληση ε, για να έρθω εδώ στη διάρκεια της συζήτησης αυτού του θέματος. Ο Αντώνιο Κώστα, ο, ο δήμαρχος της ε, Λισαβόνας, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ, έχει εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα θέματα αυτά και βασίστηκε σε έξι σημεία τα οποία θα σας μεταφέρω. Πρώτα απ' όλα, όμως ε, θα ήθελα ε, να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ε, θέλουμε έναν ενδιάμεσο στόχο ε, σε σχέση με την λευκή πίπλο. Δηλαδή, καλό είναι να πούμε ότι το 2050 θα έχουν γίνει τρομερά πράγματα, αλλά εντωμεταξύ καλό είναι να συγκλίνουμε επί ορισμένων σημείων. Πρώτα απ' πρώτο σημείο σύγκλησης, η ε, μείωση του κόστους ε, των υποδομών. Εμείς θέλουμε πλήρη εσωτερικεύση του κόστους και θα θέλαμε επίσης να δούμε εναρμονισμένη φορολόγηση σε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών. Επομένως βλέπετε ότι στην έκθεση Κώστα εμείς προχωράμε λίγο περισσότερο. Επίσης ομοφόνος πιστεύουμε ότι ε, η ε, μετάβαση από τον αυτοκινητόδρομο στην εσωτερική ε, ναυσιπλοεία και τον, το σιδηρόδρομο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο ολοκληρωτική. Θεωρούμε δηλαδή ότι ο κύριος Γκρός είναι λιγότερο επιθετικός από ότι εμείς στην Επιτροπή Περιφερειών δεν θέλει να ε, χρησιμοποιήσει ε, τον συγκεκριμένο όρο ε, «report modal», δηλαδή πλήρη μεταστροφή προς τις άλλες μορφές μεταφορών. Εμείς ζητούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημιουργίας δικτύου σταθερής τροχιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη γιατί πιστεύουμε ότι μονάχα με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει καλύτερη εδαφική και γεωγραφική συνοχή και οπωσδήποτε μικρότερο κόστος των μεταφορών αγαθών και εμπορευμάτων. Επίσης ε, θεωρούμε ότι στην δική σας ε, έκθεση ε, δεν γίνεται λόγος για την οικονομική πλευρά του θέματος, κυρίως μετά το τέλος των σημερινών οικονομικών προοπτικών. 50 δισεκατομμύρια, 50 δις ευρώ έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διάθεσή της από τα διευθυντικά ταμεία για τις μεταφορές. Επομένως εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά ε, σωστά και για υποδομές. Ε, και βεβαίως η πολιτική μεταφορών και οι δαπάνες για τις μεταφορές ε, να συνδέονται άμεσα ε, με την πολιτική ε, υποδομών αλλά και με τα διαθωτικά ταμεία. Με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορέσουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Κατά αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι τα ευρωομόλογα μπορεί να είναι μια καλή λύση για το μέλλον. Όσον αφορά τις υπόλοιπες μορφές μεταφορών, θαλάσσιες κλπ. Ε, συμφωνούμε με τον εισηγητή επίσης ε, για την αστική κινητικότητα, την κινητικότητα στις πόλεις. Ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή. Ε, θα μπορούσαμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα και να πούμε ότι θα πρέπει να ε, ε, εκπονηθεί, να δημιουργηθεί μάλλον ένα είδος βραβείου, ευρωπαϊκού βραβείου για την κινητικότητα στις πόλεις. Δηλαδή ένα είδος γαλάζιας σημαίας που θα δίνεται όχι πλέον σε παραλίες και σε θάλασσες αλλά σε πόλεις. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε λίγο την ευαισθησία Όσον αφορά την θαλάσσια κινητικότητα, ε, έχει αναφερθεί το θέμα αυτό από άλλους ομιλητές, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξαναμιλήσουμε. Ε, θεωρούμε, ε, σαν Επιτροπή Περιφερειών, ότι η πολιτική ενθάρρυνση των θαλασσίων μεταφορών θα πρέπει να είναι αποφασιστική ε, στην, ε, σε παράρτημα στη Λευκή Βίβλο ε, δεν δίνονται καθόλου ενδείξεις ότι θα ανοίξει περισσότερο κυκλοφορία στις θαλάσσιες λεωφόρους. Κυρίως όμως ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο αποφασιστικά στις ε, λεωφόρους ε, της θαλάσσης και μην ξεχνάμε ότι και εγώ ίδιος είμαι δήμαρχος της Δουκέρκης, επομένως με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Έχω πολλούς εγγεγραμμένους ομιλητές. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω να μην ξεπεράσουν τα δύο λεπτά ο καθένας για να αφήσουμε και λίγο χρόνο ομιλίας και στην Επιτροπή και στον ε, εισηγητή ε, Κατσάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έστω και αν θέματα τέτοιου είδους ε, ε, δεν μας απασχολούν κάθε μέρα ε, και μία φορά στα τόσα που έρχονται στη, για συζήτηση θα πρέπει να είχαμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε πιο ενδελεχώς. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για το μέλλον των μεταφορών, όταν μιλάμε για τη Λευκή Βίβλο, όταν μιλάμε για αυτήν την πρωτοβουλία ε, που και από τον τίτλο της καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Χάρτης πορεία για ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, φίλο Ματιό Γκρόσο που σε τέσσερις σελίδες κατάφερε ε, να συνοψίσει τα σημεία τα οποία είναι τα πιο σημαντικά και άπτονται όλων των σημαντικών θεμάτων. Το 2050 είναι ακόμα μακριά, ε, αλλά τα σημεία τα οποία έθιξε ο Ματιό Γκρός είναι πραγματικά πολύ σημαντικά. Κατά την άποψή μου, το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, λαμβάνοντα υπόψη την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη και όχι μόνον. Δεν είναι πρόβλημα μία ή δύο χωρών, είναι πρόβλημα ολόκληρη την Ευρώπη. Εμεί έχουμε 50 δι για τα δίκτυα TEN και για την ανάπτυξη των μεταφορών κατά την έννοια τη σημερινή μα συζήτηση. Όμω ο πίνακα δεν είναι πολύ θετικό. Ε, εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της οικονομίας εάν το θέλουμε και αν το πάρουμε απόφαση. Στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ακούσαμε προημερών τους, τις μεγάλες ε, ε, κεφαλές και ο Μάρκους της οικονομίας και ο Μάρκους Φέμπερ αναφέρθηκε προηγουμένως αυτό. Αλλά ακούστε, εάν σήμερα δεν κάνουμε ένα πολύ σημαντικό και αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση αυτών των ευρωομολόγων που δεν ε, ε, θα είναι μονάχα το οικονομικό τμήμα των ευρωομολόγων, δηλαδή να πάρουμε τα χρήματα και να ε, προσπαθήσουμε να κλείσουμε τρύπε των προϋπολογισμών, των κρατικών προϋπολογισμών. Εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε να μιλήσουμε για ομόλογα έργων, για project bonds που θα αφορούν σύγχρονες υποδομές εάν η Ευρώπη δεν αποκτήσει αυτές τις αποτελεσματικές υποδομές, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τότε θα έχει χάσει το παιχνίδι. Εάν ε, αναγνώσω σωστά τα όσα ακούγονται για τον εξορθολογισμό των ιδιωτικών ταμείων, για τις εγγυήσει, ε, για, για τα διάφορα άλλα προγράμματα. Μα αυτά είναι ασπιρίνες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο κακό. Εμείς σήμερα θα πρέπει να κάνουμε το πραγματικό άλμα, το πραγματικό ποιοτικό άλμα έτσι ώστε να ε, ε, βρούμε μεμονωμένα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτήσουν χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα προγράμματα υποδομών. Ο Επίτροπος, από την αρχή, ο Επίτροπος Μεταφορών από την αρχή και ο Πρόεδρος Μπαρόζο μετά ε, συμφώνησε με την εξειδικευμένη χρήση του Ταμείου Μεταφορών. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι, αφαιρε, δεν είναι έτσι αφαιρετικό και ε, ανούσιο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ απτό και συγκεκριμένο το οποίο μπορεί, εάν υπάρξει η πολιτική βούληση, να οδηγήσει σε επανεκκίνηση της οικονομίας. Και με τον τρόπο αυτό θα δοθεί συνέχεια ε, σε όλα αυτά τα οποία αναφέρονται και όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και όσον αφορά το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Γιατί διαφορετικά ε, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ευχαριστώ, ε, Καρσάνη. Κυρία Τικάου. Η ανάπτυξη του δικτύου των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σήμερα δεν είναι ισόρροπη. Η εσωτερική αγορά είναι ενιαία και απαιτεί ένα νέο μοντέλο που να προστατεύει το περιβάλλον σε όλες τις χώρες, αλλά οι συνθήκες που επικρατούν δεν είναι οι ίδιες. Επίσης τα συστήματα θα πρέπει να είναι συμβατά με εκείνα των γειτονικών χωρών. Έχουμε ε, δει τελευταία ότι υπάρχουν προβλήματα και οικονομικά. Τα κράτη-μέλη δεν τηρούν όλα ε, τις υποσχέσεις τους και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα χρειάζονται συντονισμό, αλλά χρειάζονται και χρήματα και θα πρέπει να το δουν οι μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές για να είναι βιώσιμη η χρηματοδότηση των μεταφορών. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να αναπτύξουν τα συστήματα μεταφορών τους. Δεν αρκεί το σημερινό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα και ε, τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου τα τελευταία χρόνια δεν έγινε αυτός ο εξυγχρονισμός. Γι' αυτό θα πρέπει και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσουν τον εξυγχρονισμό του υφισταμένου συστήματος και να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κράτησης ε, θέσεων για ε, τα δρομολόγια μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, τα διεθνή. Ε, ένα σύστημα λοιπόν εισιτηρίων ενιαίο ηλεκτρονικό. Και μέχρι το 2050 θα πρέπει να υπάρχει δίκτυο για τρένα υψηλής ταχύτητας που να συνδέει όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Άλλο θέμα, οι λεγόμενες θαλάσσιες λεωφόροι. Και αυτό πρέπει να το προωθήσουμε και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει σχετική πρόταση η πρόσβαση στον εύξηνο πόντο αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιείται επαρκώς, γι' αυτό πρέπει να ε, βελτιώσουμε τα συστήματα, να συνδέεται ο με το Δούναβι και τον εύξηνο πόντο. Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, θα πω κάτι που έχω επαναλάβει μέσα στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε στα νέα κράτη-μέλη νέους αυτοκινητοδρόμους Χρειάζεται παντού στήριξη και στις αστικές μεταφορές και στις περιαστικές. Και ένα τελευταίο, τα λεγόμενα ευφυή e συστήματα μεταφορών και η έρευνα που γίνεται σχετικά είναι απολύτω απαραίτητα έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές οι μεταφορές, πιο ασφαλεί. Και μιλώ εδώ για το R, ERTMS, Safe Sea Net και τα λοιπά. Χρειαζόμαστε νέα οχήματα, νέα καύσιμα και ε, νέα υποδομή και για τα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ πολύ, Λουτζάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω ε, κάτι στην ε, πρόταση του κυρίου Γκρόσο. Δεν θα ασχοληθώ με τα γενικά σημεία τα οποία έθιξε η συντονίστρια συνάδελφος Μάισνερ. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο το εξής, ε, δηλαδή μία πολύ θετική αξιολόγηση ε, για την έκθεση κυρίως στο τμήμα στο οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω ότι αυτή είναι η γραμμή που θα πρέπει να ακολουθήσει η πρότασή μας έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ε, προσδοκίες ε, τις οποίες έχουμε εκφράσει και προς την Επιτροπή όλα αυτά τα χρόνια και που θα πρέπει να ενστερνιστεί το Συμβούλιο, έστω και αν ε, έρθουμε αντιμέτωποι με αυτούς. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρξει και συγκεκριμένη αναφορά στην, για τις νησιωτικές περιοχές, στην αρχή της νησιωτικότητας. Ε, γιατί δεν αναφέρεται ε, σαφώς ε, ενώ σε αυτή την λευκή βίβλο πιστεύω ότι θα πρέπει επιτέλους να αναφερθεί η διάζουσα κατάσταση των νησιωτικών περιοχών. Ε, κύριε Πρόεδρε, μετά από δύο χρόνια εργασίας, εγώ θα εγκαταλείψω την Επιτροπή μας εδώ ε, για να πάω σε μια άλλη Επιτροπή. Δράτομαι με λοιπόν τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους, όχι μόνο του Άλντε, αλλά και όλους τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία, την ποιότητα της εργασίας μας εδώ στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ και σας αποχαιρετώ. Ευχαριστώ. Ε, ε, είναι καλό που είσαστε και μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ιζαμπέλ Ντουιρόν θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ ε, συνάδελφε για αυτήν την έκθεση και ευχαριστώ και για τα γενικά σχόλια που κάνατε προς εμένα όσον αφορά την εργασία μας εν ώψη του Συμβουλίου ε, γιατί ήμουν ήδη στην προετοιμασία του Συμβουλίου του 2001 και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να πείσει κανείς το ε, Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ συγκεκριμένοι. Ε, βεβαίως είναι γεγονός ότι δεν έχουν, και αναφέρεται στην έκθεση, ότι δεν έχουν επιτευχθεί κάποιες από τις ε, αρχές της Λευκής Βίβλου του 1 και θα πρέπει αυτά τα σημεία να καλυφθούν, αλλά δεν αρκεί ε, γιατί, τι να σας πω, ακόμα και το καλύτερη ποιότητα θερμόμετρο δεν ρίχνει τον πυρετό. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς όσον αφορά μια σειρά πραγμάτων, όσον αφορά στόχους ε, και μέσα που θα πρέπει να είναι ε, πιο φιλόδοξοι και επίσης να σημειωθεί και να υπογραμμιστεί η ανάγκη πολιτικών συμφωνιών. Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε κάποια δύναμη περαιτέρω στην έκθεση, να δούμε δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το, τον χρονικό όριο του 2020 για τις εκπομπές των, εκπομπές των αεροπλάνων ε, γιατί ε, δεν βλέπω εγώ να έχει γίνει μεγάλη πρόοδος ε, όσον αφορά ε, την ε, μείωση όσον αφορά την ε, θέση εκτός κυκλοφορίας κάποιων πολύ παλιών αεροπλάνων. Επίσης αναφερόμαστε σε μείωση 1% των εκπομπών, αλλά δεν βλέπω πώς θα επιτευχθεί αυτό, γιατί δεν βλέπω συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης, μείωση της αύξησης, μείωση συγγνώμη, του ορίου ταχύτητας, μα γιατί θα μειώνουμε την ταχύτητα ενώ διαρκώς κάνουμε πιο γρήγορα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να έχουμε και τη συνεργασία εργασία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει παρεξήγηση όσον αφορά την εξωτερήκευση του εξωτερικού κόστους, γιατί ε, κατά την άποψή μου αυτό δεν αφορά μονάχα την εφαρμογή της αρχής ε, όποιος μολύνει πληρώνει, ε, και, αλλά να υπάρξει ένας, ναι, ένας φόρος, τα έσοδα του οποίου θα δημιουργηθούν για την μείωση των, της μόλυνσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάντως είναι ε, ε, αυτή που τους αφορά αυτή η απόφαση να λαμβάνουν πάντα υπόψη τους ε, το κόστος, το περιβαλλοντικό, το ενεργειακό κτλ. Το θέμα δεν είναι να έχουμε περισσότερα χρήματα για να κάνουμε περισσότερες υποδομές. Το θέμα είναι να υπάρξουν κυρώσεις μέσα από τις οποίες θα αλλάξουν οι συμπεριφορές. Επομένως, η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους αφορά αλλαγή νοοτροπιών. νοοτροπιών. Ε, ε, ε επίσης, ε, δεν μου αρέσει η λέξη commodalité, δηλαδή πολυτροπικές μεταφορές. Ε, μου αρέσει περισσότερο στα γαλλικά η λέξη report modal, δηλαδή ε, μεταφορά προς τις συνδυασμένες μεταφορές, κίνηση προς τις συνδυασμένες μεταφορές. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης των πόλεων μας και εδώ δεν είναι πολύ φιλόδοξη η στόχη από τη μία πλευρά έχουμε ε, διπλασιασμό τουλάχιστον των ε, ε, μετακινούμενων επιβατών, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο αφορά την αύξηση των, μαζικών, το συστήματος μαζικών μεταφορών και του δικτύου μαζικών μεταφορών. Και αυτό είναι πολύ πιο φιλόδοξο. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει η σύμβαση των ε, δημάρχων είναι δηλαδή ένα δίκτυο πόλεων που δουλεύουν για την ενέργεια. Πιστεύω ότι κατά την ε, ίδια έννοια μπορούμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο ε, δημάρχων για τις μεταφορές και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα σημαία σαν την γαλάζια σημαία να είναι πράσινη σημαία όμως ο κύριος Πασκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα πω όπως μας δεσδίσατε συνοπτικά. συνοπτικά. Θεωρώ ότι σε αυτή την ε, έκθεση μπορούμε να διακρίνουμε ότι υπάρχει όπως πάντα κάνει ο συγκητής ισόρροπη αντιμετώπιση ευφυής και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι σχετικά σύντομη σε σχέση με τη Λευκή Βίβλο που είναι τόσο μεγάλη. Οπότε θα πρέπει εδώ να δούμε και να περιμένουμε ένα σωρό τροπολογίες, όχι επειδή δεν αξίζει η έκθεση, αλλά, αλλά για τέτοια θέματα συνήθως έτσι γίνεται. Οπότε θα χρειαστεί να υπάρξει κάποια συνένεση για να μπορέσουμε να διεκπεριώσουμε και να συγκεράσουμε τις διαφορετικές ε, απόψεις. Εδώ, επομένω, έχουμε να κάνουμε με μια απαρίθμηση, μια έκθεση όλων των θεμάτων που έχουν προτεραιότητα Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιολογήσουμε τα πιο σημαντικά από αυτά, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι κάποια θέματα μένουν ανοιχτά προς ε, διεκπαιρέωση. Ας πούμε, ποια είναι τα κριτήρια όσον αφορά την αναθεώρηση ε, των κανόνων που αφορούν τον χρόνο ανάπαυσης. Εδώ είχαμε πει ότι ποτέ δεν ωφελεί μια αυστηρή ρύθμιση και αντίθετα πρέπει να υπάρχει ευέλικτη αντιμετώπιση. Επίσης έχουμε τα θέματα των λιμένων ε, και κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε το τι γίνεται όσον αφορά την αναγκαία απορρίθμιση, αλλά ακριβώ θα χρειαστεί αυτή η συνδυασμένη αντιμετώπιση των μεταφορών. για αυτέ τι πολυτροπικέ μεταφορές γιατί συμφωνούμε ότι η εσωτερική του εξωτερικού κόστου των μεταφορών για όλους τους τρόπους μεταφορών είναι κάτι το οποίο διακρίνεται εδώ ότι ε, αποτελεί την απαρχή μιας συνένεση, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα, τα δίκτυα τα οποία θα υπάρχουν και δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Βέβαια ε, μιλάμε για μία Ευρώπη αλλά μία Ευρώπη με τι διαφορέ τη τις διαφοροποίησεις της. Οπότε θα πρέπει έτσι να αντιμετωπιστεί και το τι θα γίνει με ε, τα ποτάμια. Και ε, ακόμα και μέσα στην, ε, στην Ισπανία υπάρχει μεγάλη ποικιλία στη, στη, στη, στη γεωγραφία της χώρας. Ακριβώς όπως με γίνεται και με την Ελβετία. Επομένω θα πρέπει με ευφυΐα να προχωρήσουμε για να φτάσουμε σε μια τελική συνένεση, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι τα πέτυχε πάρα πολύ η ε, Κομισιόν να τα, να τα διατυπώσει όλα αυτά σε σχέση με τα όσα προσδοκούν για το μέλλον όλοι. Επομένως, μείωση εκπομπών εσωτερική εξωτερικών δαπανών, κατάργηση βαθμία των ιδιωδίων, τα νέα φιλικά στο περιβάλλον καύσιμα, αντιμετώπιση των προβλημάτων των λιμένων, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα πρέπει η Επιτροπή μας να αναζητήσει ποια είναι τα βασικότερα κριτήρια, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε κάποια έργα και προγράμματα τα οποία να είναι βιώσιμα. Επομένω, έχουμε δεδομένε τι γενικέ διατυπώσει τη Επιτροπή και εμεί θα πρέπει να προχωρήσουμε στο να τι συγκεκριμενοποιήσουμε. Επομένω, ο συγκεκριτή τα πήγε πάρα πολύ καλά, θα υπάρξουν πολλέ τροπολογίε και εγώ θα υποβάλω τι τροπολογίε. Δεν θέλω για να διορθώσω αυτά που διατύπωσε, απλώ θα πρέπει να εισφέρουμε όλοι μαζί ε, για την έκθεση. Εμεί ευχαριστούμε. Ελκαντραβή. Ευχαριστώ, πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ματιό ε, καταρχήν για το έργο του. Θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ε, τις επόμενες εβδομάδες από πλευρά της ομάδας μας. Γενικά συμφωνούμε. Το κείμενο το ίδιο είναι καλό γιατί δείχνει ε, ποιες είναι οι προτάσεις και ποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Το αρνητικό είναι ότι δεν εξηγείς αρκετά τι ε, πρόκειται να γίνει βραχυπρόθεσμα. Ε, δηλαδή το 2050 είναι πολύ μακρινό στόχος για πολλούς. Επίσης, ε, αναμένεται πάρα πολλά πράγματα από τις εσωτερικές ε, αστικές μεταφορές. αλλά εκεί η Ευρώπη δεν έχει μεγάλο λόγο. σύντομα, να σκιαγραφίσω δύο πράγματα να είναι βεβαίως πιο αηφόρο το σύστημα μεταφορών. Αυτό δεν είναι απαραίτητο μόνο για να πετύχουμε τους στόχους για το περιβάλλον, αλλά για να μην είμαστε ε, θύματα της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Είναι και ένα θέμα οικονομικό, οπότε θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος μεταφοράς. Ε, ιδιαίτερα για μεταφορές ε, πάνω από 300 χιλιόμετρα. Ε, εσωτερικές πρωτές οδοί, ε, παράκτη αναυσιπλοεία, σιδηρόδρομος, όλα αυτά τα λες, αλλά θα πρέπει να τα τονίσουμε ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται από μόνα τους. Χρειάζεται αλλαγή στην οτροπία και στη συμπεριφορά και αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις που να είναι έτσι σε λογικά οικονομικά πλαίσια και αποτελεσματικά και αποδοτικά. Και αυτό χρειάζεται επενδύσεις. Όλο το πακέτο λοιπόν που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των υποδομών ε, έχει σχέση. Ταυτόχρονα, και το θέμα το γνωρίζω πολύ καλά, θα πρέπει ε, να υπάρχουν και κίνητρα στις τιμές. Η νοοτροπία δεν αλλάζει αν, δώσεις, αν σε κάποιον ένα έναυσμα, εν πάση περιπτώσει, ε, ένα ερέθισμα. Και αυτό είναι και το θέμα της εξωτερικής, εσωτερικής του ο στόχος του 2020 για όλους τους τρόπους μεταφοράς είναι βέβαια φανταστικός, αλλά είναι πάρα πολύ φιλόδοξος αν δούμε και την οικονομική κατάσταση πώς έχει. Πάντως, ως Κοινοβούλιο πρέπει να στείλουμε όντως ένα σαφές μήνυμα για την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε. Ένα τελευταίο. Είναι βέβαια το κοινωνικό στοιχείο, έτσι και το κοινωνικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να έχουμε ενιαία αγορά μεταφορών ε, αν ε, δεν έχουμε και φιλόδοξους στόχους ε, στα κοινωνικά. Μεγαλύτερη εναρμόνιση ε, και στις αμοιβέ, καλύτερη προσέγγιση και στις συνθήκες εργασίας. Αλλιώς θα έχουμε προβλήματα απογοήτευση ματέωσης και δεν θα βρίσκουμε και καλούς υπαλλήλους. Το βρίσκουμε και μπροστά μας και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Επίσης, Μιλάς για το 2014, για την οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες. Έχεις καταλάβει ότι η ομάδα μου ε, δεν θέλει αλλαγή, δεν το θεωρεί καλή ιδέα. Είναι μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, πολιτικής για όσα πάνε στραβά στη λιμενική ε, πολιτική και στις λιμενικές υπηρεσίες. Χρειάζεται κοινωνικός διάλογος στα λιμάνια που πρόκειται να ξεκινήσει προσεχώς, θα δούμε τι θα βγει. Δεν ξέρω. Στη συνέχεια, αν χρειαστούν έξτρα μέτρα, τότε βλέπουμε. Αλλά πάντα ε, συνενετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σαΐντ. Κύριε Στσανέτσκι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, διότι μπορέσαμε όλοι μαζί να εξαγάγουμε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση και έτσι νομίζω ότι εξυπηρετούμε το σκοπό αυτό, κάτι το οποίο απαιτείτο. Τώρα, στα πλαίσια της έκθεσης Gross, θα πρέπει εδώ να σταθούμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο αποτελεί το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το ότι είμαστε ενωμένοι ε, παρά την πολυμορφία μας. Οπότε κύριε Ισηγητά, μπράβο που λάβατε υπόψη αυτή την πολυμορφία. Έχουμε αυτή την περίμετρο των 300 χιλιόμετρων, ε, κάτι το οποίο θα πρέπει και εθνικά και περιφερειακά να εφαρμοστεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ε, να λάβουμε υπόψη δηλαδή το τι ισχύει, τη διαφορά υπάρχει από το ένα μέρο στο άλλο και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Και επίση ε, μπορώ να συμφωνήσω και με την κυρία Μάισνερ όσον αφορά τι διαφοροποιήσει. Ε, διότι υπάρχουν κάποιε ε, ε δεδομένε διαφοροποιήσει όσον αφορά τον κλάδο των μεταφορών, μια που μια περιφέρεια διαφέρει πολύ από την άλλη. δεν έχουμε την περιφέρεια, την περιοχή τη Βαλτική θάλασσα που διαφέρει πάρα πολύ από την Μεσόγειο θάλασσα τελείω διαφορετικέ πραγματικότητε οπότε και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η διαφορά. Επίσης, ακούστηκαν κάποια πάρα πολύ βάσιμα επιχειρήματα σε σχέση με το πώς θα αναβαθμίσουμε τις διασυνοριακές μεταφορές, ε, κυρίως τις σιδηροδρομικές. Θεωρητικά πάρα πολύ καλά τα ακούσαμε. Πάντω να σας πω τι ισχύει στην Πολωνία. Είναι από τις πέντε φτωχότερες χώρε η Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω και θέλουμε να αναπτυχθεί η ε, διάσταση αυτή των διασυνοριακών συνδρομικών μεταφορών. Όμως εδώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τη χώρα και υπάρχει ε, συρρήγνωση των ε, συνδέσεων. Έχουμε λιγότερες διασυνδέσεις συνδρομικές και διασυνοριακές στη χώρα μας. Εντάξει για τις μεγάλες πόλεις, όμως όσον αφορά τα, τα, τα, μικρά, τα μικρότερα δίκτυα, εκεί είχαμε κατάργηση αυτών, συρρήγνωση. Οπότε παρακαλώ και αυτό να το λάβετε υπόψη στην προβληματική μας, ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας ε, κάνουμε μια ε, σύνοψη του τι ελέγχθη, διότι το ε, θέμα αυτό είναι τεράστιο, έχουμε χρονοδιαγράμματα ευρύτατα, οι επιλογές είναι περιορισμένες και επομένως ε, πάρα πολύ σωστό το πόσο ρεαλιστής ε, είναι ο συγκεκριμένο όταν μας μιλάει για την ορειβασία ε, όσον αφορά για το ότι δεν μπορεί κανείς να ανέβει απότομα στο, ξαφνικά γρήγορα στο έβρα γιατί δεν θα του λείπει το οξυγόνο άρα θα πρέπει να, προχωρήσει σιγά σιγά με, κατασκηνώνοντας στον δρόμο και έτσι θα πρέπει βαθμία να σημειώνεται η πρόοδος και ακριβώ. γι' αυτό αξίζει αυτή η έκθεση, μια που καταφέρνει με επιτυχία να συνδυάσει διαφορετικά πράγματα για αυτό το τεράστιο θέμα. Οπότε και καθήκον δικών μας είναι να διατυπώσουμε αντίστοιχα ρεαλιστικές ε, προτάσεις. Και τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη σκητάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα να Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το έργο που επετέλεσε. Ε, ήταν παράδειγμα προ μίμηση η αγαστή συνεργασία που είχαμε και επίση θα πρέπει να σα πούμε ότι για μα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το να υπάρχει αυτή η υποστήριξή σα, το ότι είμαστε εδώ στην Επιτροπή σα όλοι στο ίδιο μήκο κύματο σε σχέση και με τα όσα έχουμε πει στην ε, Λευκή Βίβλα, να σα πούμε και τι παρατηρήσει μα. Εμεί πάντω ε, ε, είμαστε πρόθυμοι προ περαιτέρω συζήτηση όμως θα θέλουμε να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη το ότι ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε τη νέα προσέγγιση. Αυτή τη διευκόλυνση για τις διευκόλυνση διασύνδεσης Ευρώπης με αυτές τις κατευθυντήριες της 10 που στις 19 Οκτωβρίου πρόκειται το TNT τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα στις ίδιες προτάσεις λοιπόν που θα κατεβάσουμε τον Οκτώβριο να το τονίσουμε όλα αυτά και ήδη είπαμε και ξαναείπαμε ότι θέλουμε να υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή για τους δρόμους στην Ευρώπη και όπως θα είπε και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής την πέσμη εβδομάδα θέλουμε να έχουμε τέτοια φιλόδοξα μέτρα του χρόνου τώρα όσον αφορά τον ενιαίο ουρανό θέλουμε ταχύτερα να προχωρήσουμε και να έχουμε ως ορίζοντα το 2013, αν δεν σημειωθεί νωρίτερα κάποιο είδου άλλη συμφωνία των κρατών μελών, επίσης πριν το χωρίσουμε στην αναθεώρηση του χρόνου οδήγηση, χρόνου ανάπαυσης του σχετικού κανονισμού, θα πρέπει να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν σήμερα, πώς μπορούμε να έχουμε πιο ομοιογενή ε, ερμηνεία, ε, ε, έλεγχο, εφαρμογή του κανονισμού ε, επίσης, ε, βεβαίω λαμβάνουμε υπόψη τους βαθυπρόθεσμους στόχους, όπως τους έχετε εσείς, για το 2020. Με κάθε επίλεξη του τι θα γίνει στο απότερο μέλλον. Πάντως, είναι δεδομένη στόχη του 2020. Για τα καύσιμα, 10% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 10% μείωση των εκπομπών, θερμοκηπίου με στόχο το 2020 και γι' αυτό θεωρούμε ο σχετική φίλος ότι έχουμε το 2050 σαν στόχους. Βέβαια, όπως θα καταλαβαίνετε, η έννοια αιτία είναι σύντομο διάστημα από πλευράς μεταφορών. Οπότε πρέπει να διαπιστώσουμε το τι γίνεται στην, ε, στις, στις αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές. Εκεί δεν προχωρήσουμε τόσο γρήγορα όσον αφορά τα βιοκαύσιμα. Ε, μια σιωπή κατά 30 των εκπομπών θεωρείται ότι είναι δύσκολο στόχο. Ακόμα και στι ε, οδικέ μεταφορέ. Η διέτηση των νέων τεχνολογιών θα είναι οριακή, μικρή. Άρα θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά το 20% προτείναμε εμείς. Και για τη μείωση επίσης, σε πρώτη φάση του 7-8% φαίνεται κάτι πιο λογικό. Κύριε Γκρός, ευχαριστούμε για τόσα είπατε για τη δική δίβλο που συμφωνούμε και επίσης εν ώψη της προετοιμασίας του προγράμματος εργασίας θα πρέπει να δούμε τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε, θα συζητήσουμε τον Νοέμβριο και έχουμε αυτέ τι ανταδράσει, της Λευκής Βίβλου να τα δούμε πώ θα τις μεταφέρουμε στην νομοθετική πρόταση Πάντως δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν νομοθετικέ λύσεις για κάθε σημείο. Είναι κατακλείδη. Θα συνεργαστούμε τόσο ώστε να φτιάξουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Πάντω ε, και τα κράτη-μέλη, οι οικονομικοί παράγοντες, οι περιφέρειε, οι χρήστε καθέκαστον είναι όλοι συνυπεύθυνοι. Είναι βέβαια και για εσά και για εμά και ένα στόχος να κινητοποιήσουμε αυτούς όλους τους ε, εμπλεκόμενου. Ήδη είχαμε τις εξελίξει στην πολιτική μεταφορών το 2001-2006, διαφορετικές φάσει και η ολοκλήρωση του χώρου μεταφορών για μας είναι ο επόμενος στόχος. Να σε ευχαριστώ, το ώστε αν, αν μπορείτε σύντομα να ολοκληρώσετε, να ολοκληρώσετε, κύριε τα μάτια. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Καταρχά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα όσα είπατε. Είμαι ήδη πεπισμένος ότι ε, θα διαμορφώσουμε μαζί το έγγραφο ε, ώστε να είναι ενδιαφέρον θα χαιρόμουν αν δεν είναι πολύ μεγάλε οι προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα. Θα επιθυμούσα να ολοκληρωθεί και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια εντός του έτους ε, ακόμα, μέσα στο 11. Αρχίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομη απάντηση. Γνωρίζω ότι ορισμένοι από τους στόχους που θέτουμε εμείς σας φαίνονται πιο φιλόδοξοι Εκεί που είναι πιο φιλόδοξη θα σας έλεγα το εξή εγώ. Με το Συμβούλιο χρειαζόμαστε συχνά ένα μικρό περιθώριο λιγμών σε πολλά σημεία. Χρησιμοποιήστε αυτή την φιλοδοξία του Κοινοβουλίου για να έχετε το περιθώριο χειρισμού απέναντι στο Συμβούλιο, αντί να μας λέτε ήδη εδώ τα επιχειρήματα του Συμβουλίου. Αυτό θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, Χαίρομαι πολύ. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν το σύστημα γενικά και θα ήθελα να απευθυνθώ στον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, Περιφερειών, στον κύριο Ντελμπάρ. Μίλησε μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη στις περιφέρειες όπου θέλουν να γίνει αυτή η αλλαγή από το ένα μέσο στο άλλο, αλλά ε, διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν χρήματα. Δεν είναι θέμα δυσπιστίας ή καχυποψίας, αλλά θέλω να προτείνω το εξή στην Επιτροπή Περιφερειών. Πρώτον, να μετρήσετε τι κάνατε για αυτά ε, με τα κονδύλια που πήρατε από τα διαρθωτικά ταμεία. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει η γνωμοδότησή σας. Πάνω από 80% πήγαν αυτά σε υποδομές αυτοκινητοδρόμων. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Δεν είναι άλλωστε του παρόντος αυτή η συζήτηση, αλλά αν κάνω μια γνωμοδότηση που ζητάει αλλαγή των μέσων μεταφοράς, δεν παίρνω τα λεφτά να τα βάλω στο αυτοκινητόδρομο. Γιατί στο παρελθόν δεν το είχα κάνει αυτό. Δηλαδή και η Επιτροπή Περιφερειών θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι με θετικό πνεύμα που το προτείνω. Να μπω και στα 300 χιλιόμετρα. Εγώ δεν θέλω να κάνουμε συζήτηση αρχής τώρα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτούμε, να δημιουργήσουμε εκείνα τα μέσα, όχι μόνο συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορεί να βοηθήσει εκεί η Επιτροπή Περιφερειών και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό. Τι κάνουμε σήμερα, ποια είναι η κατανομή στα διάφορα μέσα μεταφορά και τι στόχο έχουμε για αύριο. Θα δούμε λοιπόν τι διαφορέ από χώρα σε χώρα. Το γενικό στόχο μπορούμε πάντα να το μετρούμε, αλλά εξ όσων γνωρίζω σήμερα δεν έχουμε κανένα μέσο, ούτε περιφερειακό, ούτε πανευρωπαϊκό, που να μας λέει με μεγάλη ακρίβεια πώς έχει η κατανομή ε, ένα μέσο μεταφοράς. Αν το συζητήσουμε θα προχωρήσουμε. Για τα υπόλοιπα σχόλια, σε ό,τι αφορά το μέλλον των μεταφορών και αυτά που είπαν διάφορε πολιτικέ ομάδε. Η οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες αναφέρθηκε δις. Αυτό που με ενδιαφέρει να θυμίσω και ξέρω ότι ο προηγούμενος εισηγητής δεν έχει τις καλύτερες των εντυπώσεων, αλλά ε, η Κομισιόν είπε θα κάνουμε πρόταση. Η πρόταση μπορεί να είναι ότι δεν αλλάζουμε τίποτα και είναι εντάξει η πολιτική για τα λιμάνια. Εγώ δεν θέλω σώνει και καλά να αλλάξει αυτό ή να ε, πάει προς την ΑΒ κατεύθυνση. Απλώς δεν θέλω αύριο σε μερικά λιμάνια της Ευρώπης να λειτουργούμε και να αντιμετωπίζουμε άλλες νομικές διαδικασίες για τις λιμενικές υπηρεσίες και τη διάνοιξη των αγορών. Γι' αυτό προτιμώ να έχουμε νομοθετική παρέμβαση ή στο προσανατολισμό και στα πλαίσια του σεβασμού της ασφαλείας και γενικά της απελευθέρωσης και των ε, συνθήκων απασχόλησης εκεί. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο για τη δική σου πολιτική ομάδα, ΣΑΕΤ, για όλες τις πολιτικές ομάδες δεν μπορούμε ε, να δούμε αποκομμένη τη συζήτηση απελευθέρωσης από την ποιότητα των υπηρεσιών και από την ποιότητα των συνθηκών εργασίας ε, στα λιμάνια. σε ό,τι αφορά τα λιμάνια και πάλι και την εκπομπή των ρήπων στη θάλασσα για τη συνάδελφο Μάισναρ. Κοιτάξτε σας παρακαλώ την παράγραφο 2. Ίσως θα έπρεπε να το βάλω και στα λιμάνια, αλλά στο 2 μιλώ για τη μείωση των εκπομπών, αλλά και των άλλων ρήπων στη λαυσιπλοεία λέω, εκπομπών διοξείδου διάνθρακα και ρήπων στην αυσιπλοεία κατά 3%. Αν θέλετε να το κάνουμε πιο σαφέ. εντάξει. Για την εσωτερήκευση του κόστου, είναι εδώ η συμπατριώτησά μου από το Βέλγιο και απαντώ στα γαλλικά. Η εσωτερήκευση του χρέους δεν είναι ένα θέμα αρχή γενικά. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να το συζητήσουμε. Βεβαίω μπορεί να βελτιώσει τι υποδομέ. Δεν απαγορεύεται αυτό. Εγώ δεν θέλω να δώσω παραδείγματα για όλη την Ευρώπη, αλλά να δούμε την Ελβετία. Εγώ λέγω πάντα ότι η Ελβετία τώρα κάνει αυτό που εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε. Παίρνει χρήματα από τον ένα τρόπο και το δίνει στον άλλον αλλά το έχει βάλει στην νομοθεσία ότι θα παίρνει τα διόδια από του αυτοκινητοδρόμους για να επενδύει στο σιδηρόδρομο. Δεν λέω ότι αυτό θα είναι το μέλλον, γιατί η συζήτηση θα γίνει εμ, αβάσταχτη, αλλά μπορεί να βοηθήσει, να βελτιώσει η εσωτερική του κόστου Και αν έχουμε αύριο πιο ασφαλείς αυτοκινητοδρόμους με λιγότερα τροχεία, με νεκρούς και τραυματίες, ε, έστω θεωρώ ότι είναι σωστή επένδυση. Δεν θέλω να τα αποσυνδέσω τελείως, γνωρίζω όμως ότι ε, υπάρχει μια δυνα... Ε, δυσκολία και έχετε δίκιο για το θερμόμετρο. Αλλά εγώ θέλω να έχω θερμόμετρο για να μετράω ότι έχουμε πυρετό. Ξέρω ότι δεν ρίχνει το πυρετό, αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι έχει πυρετό. Γι' αυτό ε, πρέπει να τους πάρουμε τη θερμοκρασία έτσι από καιρό σε καιρό και αρκετά τακτικά. Συνεχίζω στα γερμανικά. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα διευρωπαϊκά δίκτυα, συμφωνούμε ότι στο μέλλον δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε τα τελευταία 15 χρόνια πολλές προτεραιότητες, ε, λίγες αναπτύξεις και παράλλαγες επενδύσεις. Νέα χρηματοδοτικά μέσα, ας μην τρέφουμε αυτά πάτες, υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα. Αλλά η ιδιωτική συμμετοχή είναι περιορισμένη, σε κάποια άλλα είναι πολύ πιο δύσκολο. Επίσης θεωρώ ότι στα μεγάλα ε, έργα θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν κάποιες παλιές ε, ε, αγκυλώσεις θα πρέπει να ξεπεραστούν. Και αυτό είναι προτεραιότητα. Δηλαδή χαρακτηρίζεται προτεραιότητα κάτι που δεν προχωράει. Δεν αμφισβητούμε καθόλου τις καλές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο συνάδελφος Πασκουάλ Ντεγκράντες ε, είπε ε, ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Τα FAPS είναι από τα καλύτερα ε, παραδείγματα και μπορεί να χρειαστούν κανένα δυο ηφαίστεια παραπάνω για να καταλάβουμε ότι ένα airblock θα ήταν καλύτερο στην Ευρώπη. Τώρα έχουμε 7. Από τα 27 γίνανε 7, το 7 στο 1 δεν χρειάζεται και τη σούπερ επένδυση. Ε, Απλώ εκχωρούνται κάποιε αρμοδιότητε και προνόμια σε κάποια κράτη. Αλλά αυτό δεν είναι εξυπηρέτηση της ασφάλειας και είναι και πιο ακριβό ε, το σύστημα σήμερα, άρα θα κάνουν και οικονομίες. Περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη οικονομία, είναι καλό παράδειγμα τα FABs. Είπα και για το σιδηρόδρομο θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα κατάλογο μη νομοθετικών πρωτοβουλειών και μη ε, ε, χρηματοδοτούμενων πρωτοβουλειών που να μην επιβαρύνουν δηλαδή τον προπολογισμό. Ζητώ συγγνώμη τώρα δεν απάντησα σε όλα όσα είπατε. Θα το κάνω σε κατηδίαν συζητήσεις που θα έχω με τους ενδιαφερομένους και εκείνους που θα κάνουν τροπολογίες. Και Πρόεδρε, παρακαλώ να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την έκθεση, για τις τροπολογίες, αλλά και για την ψήφιση στη συνέχεια. Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Τώρα είμαστε όλοι ξεκούραστοι, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, δεύτερη εν πάση περιπτώσει. Ε, μπορούμε να κάνουμε ε, τις τροπολογίες μας μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου νομίζω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Ματιέ. Η πρόταση, μάλλον το θέσω διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε πριν από το τέλος του χρόνου στην Ολομέλεια και νομίζω ότι αυτό το επιθυμούν όλοι μεταξύ των οποίων και ο εισηγητής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ήδη ψηφίσει στην Επιτροπή. Επομένως, τον Οκτώβρη θα πρέπει να έχουμε την ε, συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας επί των τροπολογιών έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την έκθεση πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει στις 12 το μεσημέρι της 20 Σεπτεμβρίου ε, να λήξει η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Είναι λίγο σύντομο το διάστημα, αλλά ε, λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις που ακούσαμε εδώ, μάλλον είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω εάν θα ε, προχωρήσουν με στη βάδα τροπολογιών. Εν πάση περιπτώσει, 20 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών, 10 και 11 Οκτωβρίου συζήτηση, ψηφοφορία 21 ε, με 23 Νοεμβρίου, σε αυτήν δηλαδή την ημερήσια διάταξη να εγγραφεί, έτσι ώστε να περάσει στην Ολομέλεια τον Δεκέμβριο του 2011. Νομίζω ότι παρότι είναι δύσκολο το χρονοδιάγραμμα, είναι ε, αποφασιστικό. Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, το οποίο είναι η δημιουργία κοινωνικού, κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας. Τόμας Ούλμερ είναι ο, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από αυτή τη συναρπαστική συζήτηση για τα μελλοντικά έργα, επανερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο ε, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 ήδη. Είναι μια συμφωνία εναέρειας κυκλοφορίας. Ο πρόεδρος διακόπτη. Μισό λεπτό, γιατί η αίθουσα αδειάζει. Παρακαλώ, αποχωρείτε ησύχως για να μπορεί να μιλήσει με την ησυχία του και με έτσι, κάποια αξιοπρέπεια ο εισηγητής. Λοιπόν, συνεχίζω. Α, σιγά σιγά αδειάζει η αίθουσα όπως είπαμε. Λοιπόν, πρόκειται για μια συμφωνία ενέργειας κυκλοφορίας της Ένωσης των κρατών μελών της και της Γεωργίας. Το Συμβούλιο έχει αποφασίσει ήδη στις 2 Δεκεμβρίου του 2010 και έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή και ήδη είναι σε εφαρμογή περιμένει τη δική μας σύμφωνη γνώμη. Δεν υπάρχουν προβλήματα μεγάλα. Η ασφάλεια, η διαφάνεια της αγοράς, της συμμετοχή στην αγορά, διαχείριση εναέρειας κυκλοφορίας, management, όλα αυτά. Δεν έχω προβλέψει τροπολογίες και περιμένω τις δικές σας προτάσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τόμας. Η κυρία Σανάλοβα. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ. πρόκειται εδώ για κάποια σημεία κλειδιά τα οποία έχει θίξει ο ε, εισηγητής και νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση μεταξύ, και ευθυγράμμιση μάλλον μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Αυτή η συμφωνία ε, μπορεί να διευρυνθεί και στην ε, Γεωργία. Βεβαίως, ε, θα υπάρξει και ενίσχυση των επαφών και, με, ε, και των υπηρεσιών μάλλον και σε πιο μικρές ε, πόλεις και με πιο μικρές ενδεχομένως εταιρείε. Η ιδιαιτερότητα της συμφωνίας με τη Γεωργία αναφέρεται σαφώς. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν περαιτέρω για τα οικονομικά και κοινωνικά περαιτέρω συστήματα. Εγώ συμφωνώ λοιπόν. Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Και για τη συμφωνία με τη Γεωργία. Όπως και στις περισσότερες άλλες συμφωνίες, είμαστε πολύ ενθουσιώδεις και υπερψηφίζουμε. Ε, εντάξει, είναι κρίμα όμως, γιατί μπορούμε να πούμε είτε ναι είτε όχι. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη θέση μας. Κατά τα άλλα, η συμφωνία αυτή είναι σε εμβρυϊκό στάδιο, είναι και μικρή. Πρόκειται για μια χώρα που είναι στην πολιτική γειτονία και θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν μιλάμε για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, καλό είναι να συνεννοούμαστε. Την ασφάλεια ε, των πτήσεων, αυτά αυξηθεί και η κυκλοφορία και οι επιβάτες. Ε, αναμένεται αύξηση 25.000 έτσι, σε πολύ ε, προσεχές διάστημα, οπότε εμεί ε, συμφωνούμε με όλα αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζιρόν θέλει να πάρει το λόγο εξ ονόματος του συναδέλφου της ή όχι. Όχι. Όχι. Εντάξει. Επομένως, Α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του σχετικά με τη συμφωνία με την Γεωργία. Πιστεύω ότι πολύ ορθώς έχουν ε, εκφραστεί ήδη τα σημεία, τα διάφορα σημεία. Να πω απλώς ε, ότι πρόκειται για μια μικρή συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα, όχι μονάχα για τη σχέση με τη Γεωργία, αλλά και με τις γειτονικές χώρες. Η λογική που ακολουθήσαμε είναι ότι θέλουμε γεωγραφική ε, σύγκληση και τεχνική συνεργασία ε, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση, μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Προσπαθούμε λοιπόν να εξεύρουμε όχι μονάχα εμπορικό ε, συμφέρον και όφελος λόγω καλύτερης πρόσβασης ε, και ε, στην αγορά, ε, για λόγους τουρισμού ή ή εμπορικών πούμε, συμφωνιών, αλλά ε, και ε, μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης θεωρούμε ότι είναι ένα καλό πρώτο βήμα για να διευρυνθούν ε, οι συμφωνίες αεροπορικού χώρου και με γειτονικές χώρες. Και μάλιστα βλέπω ότι μετά αναφέρεστε στο ημερήσιο πρόγραμμά σας και στην Ιορδανία Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πιο συνολικό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρο. Ο εισηγητή θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένως, υπενθυμίζω ότι μπορούν να υπάρξουν ε, τροπολογίες επί, επί του σχεδίου έκθεσης, ε, όχι όμως επί του αρχικού ε, ε, κειμένου και επομένως το Νοέμβριο 2011 στην Ολομέλεια θα γίνει η ε, ψηφοφορία. Φτάνουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας για τις ε, αεροπορικές μεταφορές, η κυρία Σεναλόβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι με αυτή τη συμφωνία ε, προχωρούμε σε μια νέα κατάσταση. Πριν το 2008 ήταν διμερείς οι συμφωνίες και τώρα ε, είναι μια ε, συνολική συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές αντικαθιστά τις προηγούμενες διμερείς συμφωνίες και έχουμε μια ενιαία προσέγγιση. Τρεις είναι οι στόχοι μας εδώ. Η σταδιακή διάνοιξη της αγοράς ε, για τα δρομολόγια, για την πρόσβαση και για τις δυνατότητες, μη διάκριση, ε, ίση όρη ανταγωνισμού με βάση των αρχών των συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνθήκων και Επίσης θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι προδιαγραφές της Ιορδανίας στους διάφορους τομείς στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται και στον εξυγχρονισμό της Ιορδανικής οικονομίας. Μετά τη Σαουδική Αραβία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο παριθμόν ένα εμπορικό εταίρος της Ιορδανίας. Η, η συμφωνία αυτή είναι λοιπόν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικό στοιχείο της πολιτικής γειτονίας σύμφωνα με εκτιμήσεις ε, ε, που βγήκαν από εξωτερική μελέτη που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αυξηθούν οι επιβάτες κατά 54.000 και ε, οι καταναλωτές που μπορούν να επεφελούνται μέχρι 30 εκατομμύρια. Υπάρχει δυνατότητα να διευρυνθεί αυτή η συμφωνία και σε άλλες χώρες της Μεσογείου και να έχουμε μια ενιαία συμφωνία και νέο χώρο. Θεωρώ ότι αυτό είναι στο, προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάδει με την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και... Πρόεδρε, ήθελα να σας πω μόνο συμφωνούμε με την πρόταση αυτή και με την έκθεση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το ΕΛΚ. Το υποστηρίζουμε ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θεωρώ θα πρέπει να συμφωνήσουμε ε, απολύτως. Ε, πάντα συγκρίνω τι συμφωνίες, οι οποίες βέβαια διαφέρουν μεταξύ τους, για την Ιορδανία σε σχέση με τη Γεωργία. Δεν είναι πιθανή μελλοντική χώρα της Ένωσης, διαφορετικό, παρόλα αυτά σημαντικό. Κάτι άλλο που μου αρέσει πολύ είναι και η μελλοντική διεύρυνση σε μια κοινή συμφωνία με υπόλοιπε χώρε τη Μεσογείου γενικώ, διότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Και όπως είπατε, σε πρώτη φάση θα έχουμε ε, και περισσότερους επιβάτες και περισσότερα πλέον εκτήματα, πρόσβαση μεγαλύτερη. Συμφωνούμε κι εμείς. Ευχαριστώ και την κυρία Σενιάλοβα για την έκθεσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σνέρε. Ε, κυρία Ντυρό, βεβαίως ως πράσινοι εμείς ε, θα υπερψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. όμως ε, πρέπει να πω ότι η συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε πριν αρχίσουν ε, οι διάφορες ταραχές ε, πρέπει να πούμε ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες σε αυτή την πλευρά, σε αυτή τη γεωγραφική περιφέρεια θα πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούν στην δημοκρατική μετάβαση των χωρών αυτών. Απλώς ήθελα να σημειώσω ότι έχει αλλάξει τελείως πλέον ε, που είμαστε υποχρεωμένοι με την καλή έννοια το λέω να δουλέψουμε το νέο λοιπόν πλαίσιο ε, το οποίο θα μας οδηγήσει και σε κάποιες διαφορετικές ενδεχομένως θεωρήσεις. Ευχαριστώ πολύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, ε, για την εισηγήτρια μάλλον, για το σχέδιο έκθεσης, το οποίο υπέβαλε και το οποίο ενστερνίζεται πλήρως τις αρχές της ε, πρότασης ε, ε, είναι σημαντικό το σημείο το οποίο έθιξε η κυρία Μέσνερ, δηλαδή ότι η Ορδανία δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κράτος μέλος, επομένως υπάρχουν κάποιες διαφορετικές αποχρώσεις σε σχέση με τη Γεωργία. Τούτου λεχθέντος πάντως πρέπει να πούμε ότι ειδικά αυτή η συμφωνία με την Ιορδανία εγγράφεται σε μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, ε, γιατί εμείς είχαμε κάνει πολλές δραστηριότητες και πολλές κινήσεις όσον αφορά την πρόθεση των αερομεταφορών πριν από το κείμενο αυτό ε, και πρέπει να πω ότι το σύνολο ας πούμε ε, των προγραμμάτων ασφαλείας ε, της Ιορδανίας είναι απολύτως συμβατά και άλλωστε έχουν εμπνευστεί από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και σε άλλους τομείς συνεχίζουμε την εργασία και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι την ανάλυση της κυρίας Ντυρόν, δηλαδή ότι υπάρχει ε, ε, ένα, μια ευτυχής αλλαγή ε, πλαισίου που οπωσδήποτε θα παίξει κάποιο ρόλο. Ενδεχομένω λοιπόν οι συμφωνίες αυτές θα έχουν μια ακόμα μεγαλύτερη έννοια γιατί θα αφορούν το άνοιγμα της Ευρώπης προς τις χώρες αυτές, αλλά ενδεχομένως και άνοιγμα των χωρών αυτών ε, της μίας προς την άλλη μεταξύ τους. Ε, και οπωσδήποτε θα ακολουθηθεί και από άλλες ε, συμφωνίες με το Μαρόκο. Ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσουν διεργασίες με την Τινησία και επομένως προσέγγιση της Ευρώπης με τις χώρες αυτές, αλλά και προσέγγιση των χωρών αυτών μεταξύ τους. Ευχαριστώ λοιπόν την Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την ε, έκθεση ε, αυτή και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μήπως ε, η συνάδελφος Σενάλοβα θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι. Μπορούν να υπάρξουν λοιπόν τροπολογίες επί του νομοθετικού ψηφίσματος αλλά όχι επί της ιδίας της συμφωνίας. 20 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία υποβολής τροπολογιών, ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών τον Οκτώβριο και Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι ο Ματιέ θα μας πει δυο λόγια τώρα για την επόμενη έκθεση που αφορά την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και ο Μάριαν Μαρινέσκου δεν είναι εδώ. Ακριβώς κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Μαρινέσκου δυσκολίεται και που και με παρακάλεσε να σας παρουσιάσω σύντομα τη γνωμοθέτηση του, τη έκθεση για το 2010, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και τους διάφορους τομείς, τη διαφάνεια, το κόστος, τα τέλη, στο σιδηρόδρομο, γιατί είμαστε μεσούς της συζητήσεως, δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό ε, που βλέπουμε στα διάφορα θέματα περαιτέρω διάνοιξη δηλαδή των σιδηροδρόμων και ένας ενιαίος σιδηροδρομικός χώρος, η ε, ανεξαρτησία των παρόχων υπηρεσιών από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ε, ενίσχυση του, της ρυθμιστικής αρχής, αλλά κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι τα χρέη των σιδηροδρόμων, των ιστορικών ε, σιδηροδρομικών ε, οργανισμών των διαφόρων κρατών. Από χώρο σε χώρο διαφέρει πάρα πολύ η κατάσταση στο παρελθόν. Ε, ήταν διαφορετική η κατάσταση. Είχαμε ουσιαστική πλήρη παραγραφή του χρέους μερική ή ενδεχόμενη. Δεν είναι ένα θέμα που στερείται ενδιαφέροντος. Καλό θα ήταν να το κοιτάξουμε κι εμείς έτσι σε μεγαλύτερο βάθος και λεπτομέρειες. Μεταξύ άλλων αυτό ξεκαθαρίζει και τη στάση ορισμένων κρατών μελών όταν πρόκειται για τη συνεργασία ε, παρόχου υπηρεσιών και συντηροδρομικής επιχείρησης, γιατί συνδέεται και με ένα άχθος από το παρελθόν, ένα βάρος του χρέους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Επίσης γίνεται λόγος για τις αερομεταφορές που θα μας απασχολήσουν στο προσεχές μέλλον, κυρίως για τα λεγόμενα σλότς, τις χρονοθυρίδες και τον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό και κάτι άλλο που επίσης έχει ενδιαφέρον, υποστήριξη των ε, αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους. Είχαμε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντίστοιχες τοποθετήσεις του παρελθόν. Ε, Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις ε, διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης για να προσελκύσουν αυτές τις εταιρείες, μεταξύ αυτών και στη χώρα μου. Στις θαλάσσιες μεταφορές, ε, χρηματοδότηση των υποδομών των θαλάσσιων λιμένων για τον εξυγχρονισμό. Αυτό θα μπορούσε να συντηθεί σε ένα πακέτο για τις λιμενικές υπηρεσίες. Τι ε, μπορεί να γίνει στο μέλλον. Πάντως νομίζω ότι έχει σημασία να αξιολογήσουμε για αυτά τα στοιχεία με μεγαλύτερη ακρίβεια για να δούμε τι γίνεται και στην έκθεση ανταγωνισμού, ποια είναι τα βασικά δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα των επιβατών. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ ε, ο κύριος Μαρινέσκου να υπάρχει ένα εγχειρίδιο, ένας οδηγός για τους επιβάτες. Ε, εδώ έρχεται να προσθεθεί και ο κλάδος του τουρισμού για τη διαφάνεια, για την ενημέρωση, για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των τουριστών. Είναι πρόσφατη η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και ακόμα σε εμβρικό στάδιο Λοιπόν, η διάνοιξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το έχουμε συζητήσει αυτό, τώρα τι γίνεται με την εφαρμογή. Τα ξέρουμε αυτά. Και αυτά. Σε ορισμένε χώρες και περιφέρειες χρειάζεται επιτάχυνση. Και κατά την άποψή μου, θα μας απασχολήσει και στην Επιτροπή μας στο μέλλον η αξιολόγηση. Αυτονόητο και προφανές. Αυτά είχε να σας πει ο κύριος Μαρινέσκου για την έκθεση του, την γνωμοδότηση μάλλον. Ε. Ευχαριστώ πολύ Ματιέ, ο Σαΐντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε και μπορούμε να τον ακολουθήσουμε, αλλά θεωρούμε ότι η γνωμοδότηση αυτή το παρακάνει από ενθουσιασμό στην απελευθέρωση. Δεν είναι πανάκια ούτε για ε, το σιδηρόδρομο ούτε για το ταχυδρομείο ε, την οδηγία αυτή και δεν αναφέρεται ε, πολύ συγκεκριμένα της Υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Και σε αυτά τα θέματα ε, για τις υπηρεσίες, για τις υπαροχές και τις συμβάσεις θα κάνουμε τροπολογίες να βελτιώσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ Σαΐτ, ο κύριος Δεμπάκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Στην παρθενική μου ομιλία, σε αυτή τη φοβερή σας επιτροπή, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση, αλλά δεν περίμενα ε, τίποτα διαφορετικό. Ξέρετε ότι έχουμε και εμείς τροπολογίες και παρατηρήσεις. Η εσωτερική αγορά για να ολοκληρωθεί ε, έχει ένα βασικό στοιχείο που είναι η ολοκλήρωση και των μεταφορών. Και ζητάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τις κρατικές ενισχύσεις, τις άμεσες όμως και έμεσες για τις υποδομές και τη χρηματοδότησή τους ε, ήδη από σήμερα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις μεταφορές, αλλά και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες από ό,τι κατάλαβα. Επιπλέον, ε, τον ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν είναι θέμα μόνο της Επιτροπής, αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων και γρήγορα να φέρουν αντίστοιχες προτάσεις, Έχουμε και τις αποφάσεις του δικαστηρίου ε, για την απελευθέρωση των επιβατικών μεταφορών. Χρειάζονται να γίνουν ακόμα μεγάλα βήματα. Η αναδιατύπωση της οδηγίας, το recast, έχουν γίνει μεγάλες συζητήσεις. Ε, θα πρέπει το κείμενο να είναι ε, σε συνάφεια και συνοχή με το προηγούμενο, να είναι πραγματικά ανεξάρτητη η αξιολόγηση και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αεροπορικές εταιρείε και τις νέες χρονοαφυρίδες. Ε, θα δούμε τι ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάλι η διαφάνεια πρέπει να κυριαρχεί. Ο κώδικας για τα δικαιώματα των επιβατών, αυτό έχει σημασία για όλα τα μέσα μεταφοράς, να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους, αλλά να συντονίζονται και καλύτερα. Μια εγκάρσια λοιπόν οριζόντια προσέγγιση χρειάζεται ε, οπωσδήποτε. Σύντομα και για την υποδομή των λιμένων, των θαλασσίων, είναι πολύ σημαντικό αυτό και παραμένει να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια για τη χρηματοδότηση των ε, λιμενικών υποδομών και απελευθέρωση και διαφάνεια στην απελευθέρωση. Και ένα τελευταίο, δικές μεταφορές. Ο εισηγητής δεν λέει σχεδόν τίποτα στην γνωμοδότησή του για αυτές αλλά θα ήθελα εγώ να τονίσω ότι ισχύουν νέοι κανόνες τώρα για ε, το καμποτάζ, για την εσωτερική, μάλλον ενιαία αγορά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να απελευθερωθεί η αγορά μας, να ανοίξει περισσότερο για να λειτουργεί καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, εμείς βέβαια και συμφωνούμε με αυτούς τους στόχους για την ε, διαφάνεια, για την ε, άμεση και έμεση εξοικονόμηση δαπανών. Είναι βασικό αυτό και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά καθορισμένο και τώρα έχουμε για τις αεροπορικές μεταφορές στο σημείο 9. Θεωρούμε ότι θα πρέπει και αυτό να το κάνουμε έτσι ώστε για τις ολικές υπηρεσίες, καθολικές υπηρεσίες. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για αυτό το στόχο, γιατί θα πρέπει αυτό να καλύψει τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν διάφορες παροχές ε, που παρέχονται από τις εταιρείες, όμως αυτό δεν δικαιολογεί το εξωτερικό ούτε το εσωτερικό ε, κόστος. Και έχουμε επομένως κάποιες φοροαπαλλαγές, οι οποίες πλέον εδώ τις καταγγέλουμε, δεν είναι πια αποδεκτές, είναι, είναι είναι άδικες. Όμως θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ε, υποστήριξη του δημοσίου τομέα χρειάζεται μια προσεκτική προσέγγιση με την απορρίθμιση να θέλουμε να αποφύγουμε την ε, απόλυτη διάλυση της ε, λειτουργίας των υπηρεσιών σε δίκτυο επομένω ακριβώς όσον αφορά τους σιδηροδρόμους θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ιστορικούς παρόχους οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και επομένω ε, θα πρέπει να μην ε, οδηγηθούμε σε κάποιο είδου αποδιοργάνωση και αυτό θα είναι επιδείνωση της καταστάσεως. Επίσης θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα να σκεφτούμε κατά πόσο μπορούμε να ξαναδώσουμε κάποιο είδου ε, ενισχύσει για την ισοδρομική μεταφορά των εμπορευμάτων και θα πρέπει κάποιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτός ανταγωνισμός. Είναι πολύ ε, συγκεκριμένος αυτός ο κλάδος. Και θα πρέπει και εδώ να δούμε πώς εδώ να έχουμε κρατική ενίσχυση για να μπορεί να γίνει η δουλειά. Σας ευχαριστούμε. Πριν το στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας πω δύο λόγια όσον αφορά αυτό το, αυτή την έκθεση στον τον ανταγωνισμό, διότι τελικά μιλούμε περισσότερο για αυτού του είδου ε, τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφορά, ε, ούτως ώστε να κινούμε προς σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά βέβαια, ε, είναι άλλο, άλλο, είναι άλλος τομέας ο ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται συγκεκριμένο πρόβλημα των ε, μεταφορών και αποτελεί μια άλλη προβληματική. Καλή κακή τρόπο μεταφοράς, οικολογική τρόπο μεταφοράς, η εξοικονόμηση δαπανών. Κάτι το οποίο με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι διαπιστώνουμε ότι είναι δυνατόν ε, μπορεί κανεί να κάνει τη μεταφορά με πολλούς τρόπους, οπότε τελικά αναδύονται τα ίδια και τα ίδια προβλήματα που αφορούν κάθε μέθοδο μεταφοράς, κάθε τρόπο μεταφοράς. Αυτά τα προβλήματα, τα τα γνωστά. Έχετε το λόγο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρσι δουλέψαμε πάρα πολύ εντατικά όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την εφαρμογή του δικαίου και αυτό φαίνεται και στην κρίση. Χαιρετίζουμε την έκθεση Μαρινέσκου. Δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο σε αυτή τη φάση να παρατηρήσουμε. Λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που βεβαίως τις γνωρίζουμε ήδη και θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις πρώτα από το ιστοσημείο υπαριθμών 2 όσον αφορά την διαφάνεια για κόστος, ε, τις διαφορετικές δαπάνες, γιατί ο κλάδος αυτό προσδοκά, περισσότερη διαφάνεια. Όπως έχει σήμερα το δίκαιο, δεν απαιτεί τα κράτη-μέλη να κοινοποιούν τα δεδομένα σχετικά με τις ενισχύσεις. Ε, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν, δεν έχει τα, τα στοιχεία αυτά τα απαραίτητα για να το ελέγξει αυτό. Τώρα όσον αφορά τις ακυρώσεις έχουμε τις κρατικές ενισχύσεις για δομικέ μεταφορές. Τα λέμε στο κεφάλαιο 4 και εδώ προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες για ακυρώσεις, ματαιώσεις. Ε, προς το παρόν δεν προβλέπεται να κάνουμε κάποια αλλαγή σε αυτή τη ρύθμιση και όσον αφορά τις υποδομές στα λιμάνια. Έχουμε κάποια μελή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα ολοκληρωθεί και θα δώσει αποτελέσματα αρχάς 2012, οπότε θα αναλύσουμε προσχετικά και τα δικά σας τα στοιχεία και επί τη βάση των μελετών της δικής μας και της δικής σας θα συνεχίσουμε το έργο μας και τις αμέσως επόμενες εβδομάδες περιμένουμε πώς και πώς να το ξανασυζητήσουμε μαζί σας. Ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρο. Ματιέ, θες κάτι να προσθέσεις. Ε, θα τα διαβιβάσω αυτά στον εισηγητή, όπως καταλαβαίνετε, στον κύριο Μαρινέσκο και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ελπίσουμε ότι παρά τις διαρθρωτικές αλλαγές στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση MOVE, θα ε, υπάρχει συνεργασία μεταξύ ανταγωνισμού και μεταφορών, γιατί οι μεταφορές έχουν και τις ιδιαιτερότητέ τους που θέλουμε και εμεί στην Επιτροπή μας εδώ να λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ίδια προθεσμία υποβολή τροπολογιών 20 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας τον Οκτώβρη. Να ξέρετε ότι η αρμόδια επί της ουσίας είναι η οικονομική και θα ψηφίσει στις 22 Νοεμβρίου και ενδεχομένω θα προλάβουμε να ε, το, περάσουμε το θέμα στην Ολομέλεια, στην τελευταία Ολομέλεια του χρόνου. Δεν έχουμε τίποτα ήποτα διάφορα και ολοκληρώνουμε λοιπόν τις εργασίες μας ε, λίγο νωρίτερα. Θα τα ξαναπούμε στις 10 Οκτωβρίου στις 3 το απόγευμα στις Βρυξέλλες.